Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην Υποεπιτροπή, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλώς ορίζουμε όλα τα μέλη της Υποεπιτροπής και τους προσκεκλημένους. Θα συνεχίσω στην πολωνική γλώσσα την ομιλία μου. Έχετε λάβει όλοι την ημερήσια διάταξη για σήμερα. Υπάρχουν σχόλια επί της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ας περάσουμε στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης ε, της ανακοινώσεις του Προέδρου. Πρώτα απ' όλα έχω κάποια καλά νέα να μοιραστώ μαζί σας από τις Ηνωμένες Πολιτείες άλλη μία πολιτεία. Το Connecticut ανακοίνωσε ότι πρόκειται να καταργήσει τη θανατική ποινή. Πρόκειται για τη 17η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών που καταργεί τη θανατική ποινή και την πέμπτη εντός ε, πέντε ετών που πραγματοποιεί μια τέτοια κατάργηση. Ο κυβερνήτης κ. Μαλόη υπέγραψε το νομοσχέδιο την περασμένη Τετάρτη, το οποίο τεθεί σε ισχύ αμέσω, αλλά δεν είναι αναδρομικό. Ισχύει μόνο για το μέλλον. Ταυτόχρονα η θανατική ποινή θα αντικατασταθεί από την ισόβια κάθερξη. Αυτό θα ισχύσει μόνο για μελλοντικές υποθέσεις. Θα ήθελα επίσης να μοιραστώ μαζί σας μερικές πληροφορίες ε, σχετικά με τον Νότιο Σουδάν. Οι διανέξεις ε, συνεχίζονται στα σύνορα μεταξύ Σουδάν και Νοτιού Σουδάν. Η περιοχή που πλήττεται περισσότερα είναι τα βουνά Νιούμπον στην νότια πλευρά ο αριθμός μεταναστών που αναζητούν καταφύγιο πέρα από τα σύνορα του Νοτιού Σουδάν αυξάνεται καθημερινά και σήμερα έχουμε πάνω από 23.000 πρόσφυγες ε, στο στρατόπεδο Ίντα. Αυτό μπορεί να κλιμακωθεί σε σημαντική ανθρωπιστική κρίση, ε, ιδιαίτερα δεδομένου ότι ξεκινάει σύντομα η εποχή των βρεχών, που σημαίνει ότι θα υπάρχει δυσκολία παροχής των βασικών ειδών και τροφίμων σε αυτούς τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων, ε, του των Εθνών ε, υιοθέτησε ένα ψήφισμα που απειλεί κυρώσεις και προς τις δύο χώρες εάν δεν διακοπεί η κλιμάκωση και αν δεν ξεκινήσουν συνομιλίες εντός δύο εβδομάδων μεταξύ των δύο μερών που θα πρέπει να καλύψουν ε, τόσο τα έσοδα από το πετρέλαιο όσο και την οριοθέτηση των συνόρων με έναν τρόπο ειρηνικό βασισμένο σε συμβιβασμό τα σύνορα μεταξύ αυτών των δύο χωρών αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα διακυβεύματα όσον αφορά τις αμοιβέ ε, σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο χωρών. Τρίτον, θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω και για ένα άλλο θέμα. Άλλη μία απεργία πείνας ε, Παλαιστινίων έχει ξεκινήσει. Ο ε, ο πρόεδρο της ε, Επιτροπής έχει ενημερωθεί από τον κύριο Γιάκομπι Κλώτ, συντονιστή της ε, εκστρατεία Open the Doors. Πρόκειται για έναν οργανισμό που συγκεντρώνει 410 βουλευτέ από τα 27 κράτη-μέλη και οι πληροφορίε που διαβιβάστηκαν ήταν για δύο Παλαιστίνιους ε, κρατούμενους που βρίσκονται στην 72η ημέρα της απεργίας πείνας τους και αν συνεχίσουν αυτή την απεργία πείνας ε, οι ζωές τους θα κινδυνεύσουν. Εκτός από αυτούς τους δύο υπάρχουν και πολλοί άλλοι κρατούμενοι σε απεργία πείνας εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε επίσης άλλους, άλλα 2.000 άτομα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες που κάνουν απεργία πίνε Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε λάβει κάποιε πληροφορίε σε σχέση με τις συνθήκες κράτηση. Ε, πληροφορίες ε, για ευτελιστική και ε, αντιμετώπιση, σωματική έρευνα των επισκεπτών, μη ε, σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων των επισκεπτών. Για παράδειγμα, δεν τους επιτρέπουν να συνεχίσουν την εκπαίδευση, ζήτημα το οποίο επεσήμανε ο κ. Γιάσο. Ας περάσουμε τέταρτον στην Ιεμένη. Η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον κ. Λογμπελέρ και με τη συνοδεία του κ. Χάουρτ και Πρέδα επέστρεψε από την Ιεμένη χθε, εάν δεν κάνω λάθος. Κατά την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας θα ακούσουμε μια πλήρη έκθεση σε σχέση με αυτή την επίσκεψη. Η κυρία Λόγκουερα θα βρίσκεται εδώ αργότερα σήμερα και θα συνεχίσει να προεδρεύει την ε, συνεδρίαση ήρθε αργά από την Ιεμένη χθε. Στον Μπαχρέν και άλλα ζητήματα στι 29 Απριλίου η συνάδελφο Άννα Γκόμε προσγειώθηκε στη Μανάμα, αλλά δεν τη επιτράπηκε να εισελθεί στη χώρα. Δεν τη επιτράπηκε να επισκεφθεί τη χώρα. Τη ζητήθηκε να εξηγήσει γιατί ήθελε να επισκεφθεί τη χώρα και τη ζήτησα σαν να παρέχει τα στοιχεία επικοινωνία των ατόμων που θα επισκεπτόταν. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι συστήθηκε ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έδειξε το πορτογαλικό διπλωματικό διαβατήριο πέντε ώρες αργότερα δεν είχε ληφθεί απόφαση. Δεν της επετράπη να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν ζήτησε την άδεια να επισκεφθεί την Δανέζα ακτιβίστρια ζήτησε το τηλέφωνο της ε, και το τηλέφωνο του ε, κ. Τζίση, δικηγόρου. Ζήτησε επίσης να επικοινωνήσει με τις ε, αρχές του Μπαχρέιν ώστε να λάβει πληροφορίες σε σχέση με τον Αμπελάχη Αλκαβάγια, πατέρα της, που πρόκειται για ενεργό ακτιβιστή ο οποίος ε, έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη λόγω της συμμετοχής του σε ε, διαδήλωση κατά της κυβέρνησης το περασμένο έτος. Κατά τη διαμαρτυρία του ξεκίνησε μια ανοιχτή απεργία πείνας πριν από πάνω από 82 μέρες. Ε, πέρασαν 7 ώρες, αλλά οι αρχές του Μπαχρέιν αρνούνταν στην κυρία Γκόμες τη θεώρηση εισόδου και ζήτησαν να εγκαταλείψει τη χώρα. Η πρόεδρός μας ε, έγραψε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρεσβευτή του Μπαχρέιν, ο κύριος Σούλτς, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης απευθύνθηκε στις αρχές του Μπαχρέιν για το ίδιο ζήτημα. Θα πρέπει επίσης να προσθεθεί ότι μια ομάδα του BBC επισκέφθηκε τον κύριο Αλκαβάια στο στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μπαχρέιν. Αυτή η επίσκεψη έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα. Ο κύριος Αλκαβάια δήλωσε ότι είχε καλή μεταχείριση στο νοσοκομείο ε, με εξαίρεση την ε, ξαναγκαστική διατροφή του, την οποία αρνείται το νοσοκομείο. Την ημέρα πριν από την επίσκεψη, η ομάδα δικαστών αποφάσισε ότι αυτή η υπόθεση και οι υποθέσεις 19 άλλων αντιφρονούντων δεν θα ε, δικάζονταν από στρατιωτικό αλλά από πολιτικό δικαστήριο. Α περάσω τώρα στην ακρόαση του Βεράσουν Ντούμα. Στην τελευταία διευρυμένη συνεδρίαση του Προεδρείου της ε, Υπεπιτροπής Ντροάη, η κυρία Πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι θα γίνει μια ακρόαση στη Μόσχα υπό την Προεδρία της Ρωσικής Δούμας που αφορά τις παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην, ανθρώπινη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περασμένη εβδομάδα η κυρία Πρόεδρο ε, έλαβε τη σχετική πρόσκληση που μας καλεί να συμμετέχουμε στην προανεφερθήσα ακρόαση. Η κυρία Λόγχ ε, Μπίλερ ε, αρνήθηκε την πρόσκληση. Ταυτόχρονα έλαβε και ο Σμπλοκ την ίδια πρόσκληση και διαβίβασε το σχετικό σημείωμα στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στη Μόσχα που θα συμμετέχει ως παρατηρητή σε αυτή την ακρόαση. Βερμανία. Οι τελευταίες εκλογές ε, του Απριλίου και η αβεβαιότητα πριν από τις εκλογές για το κατά πόσο η Άντσαν Σουτσί και το κόμμα της θα λάμβαναν έδρα στο Κοινοβούλιο λόγω της ε, ανάγκης διασφάλισης του συντάγματος ε, το οποίο σύνταγμα είναι αμφίβολο κατά πόσο είναι δημοκρατικό. Ο, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη μπορούμε τώρα να πούμε ότι είμαστε βέβαιοι ότι τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου θα λάβουν τις έδρες τους στο Κοινοβούλιο. καθώς αποδέχθηκαν ότι θα σέβονται το Σύνταγμα, το Σύνταγμα το οποίο μας προκαλεί ισχυρές αμφιβολίες σε εμά εδώ στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βερμανία. Οι περισσότερες ε, κυρώσεις έχουν ανασταλεί εκτός από το εμπαργό όπλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει το γραφείο της στη Βερμανία γεγονός που θα μπορεί να μας δώσει μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της κατάστασης και θα μας δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε ενημερωμένες πληροφορίες όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση και τις πολιτικές εξελίξεις στη Βερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βεβαίω με το βραβείο Σαχάροφ θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ενεργά. Πρόκειται για ε, μείζονο σημασία ε, ε, ένδειξη για το ε, ρόλο που θα παίξει το κόμμα της Άγκσαν Σούση στη Βερμανία. Τώρα η Κίνα, η περίπτωση του Τσέν Τσέγκ, τα μέσα ανέφεραν ευρέως για τον ακτιβιστή Τσαν Κουάν που διέφυγε από την κατοικοκράτηση και διέφυγε στην ε, Αμερικανική Πρεσβεία στο Πεκίνο. Αυτή η υπόθεση δείχνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν δευτερεύουσα σημασία ζήτημα αλλά ζωτικό ζήτημα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Το κοινοβούλιο μας ε, έχει αρχίσει να εξετάζει αυτό το θέμα ήδη από το 2006 όταν ο εν λόγω ε, πολίτης ε, καταδικάστηκε σε φυλάκιση μετά από την έλλειψη αντίδραση της Κίνας ε, για το σύντομο διάστημα στο οποίο παρέμεινε στην πρεσβεία ο κ. Τσάν αρχικά επιθυμούσε να παραμείνει στην Κίνα επικρατούσε το γεγονό ότι θα υπήρχε σεβασμό των δικαιωμάτων του. Μετά όμω έκανε αίτηση να φύγει από την Κίνα μαζί με την κυρία Κλίντον στο ίδιο αεροπλάνο. Έλαβε κάποιε ενδείξει τόσο από τι ΗΠΑ όσο και από την Κίνα ότι θα το επιτρεπόταν να αναχωρήσει από την Κίνα ως ε, υποψήφιος φοιτητής που θα συνέχιζε τις σπουδές του στις ΗΠΑ. Οι Κινέζικες αρχές υπενηχθήκαν ότι η προϋπόθεση θα ήταν να ε, διαθέτει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και ότι σε αυτή την περίπτωση το καθεστώς φοιτητή θα αποτελούσε, θα αποτελούσε ικανή συνθήκη για να λάβει το, την άδεια να ταξιδέψει. Αυτή τη στιγμή το ζήτημα που ανακύπτει είναι το εξής. είπατε εκπρόσωπο Λέδη δηλαδή, Αστόρ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι πρόκειται να κάνουν όταν θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα γεγονότα που αφορούν αυτόν τον συγκεκριμένο Κινέζο αντιφρονούντα. Θα καταλήξουν σε άλλη μια σειρά από κυρώσεις ε, επιβάλλονται στις περιπτώσεις ε, Κινέζων αντιφρονούντων που καταφεύγουν σε δυτικές πρεσβείες. Ο κύριος Τσάνγκουαν Τσάνγκα παραμένει απομονωμένο σε ένα νοσοκομείο στο Πεκίνο αναμένοντα νέα όσον αφορά τη μοίρα του. Δυστυχώ κάποιοι από του φίλου και του συγγενεί του που ενεπλάξαν στη διαφυγή του έχουν εξαφανιστεί και ενδέχεται να έχουν αντιμετωπίσουν σοβαρέ συνέπειε. Θεωρούμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ελευθερία και τα βασικά δικαιώματα του κ. Τσανκουάνγκ δεδομένης της ε, ε, μακροχρόνιας καταδίκης τους και της παρανομής κατοίκων ε, κράτησής του. Τόσο και τον κύριο Γκουαντζέγκ όσο και την οικογένειά του θα πρέπει να ε, απολαύσουν τα βασικές τους ελευθερίες. Επίσης έχουμε ενημερωθεί ότι η αστυνομία ανέκρινε επίσης τον Χουιάρ τον βραβευμένο με το βραβείο Σαχάροφ και κοντινό φίλο του κυρίου Κουαντσέγγ. Αυτέ ήταν οι πληροφορίε που ήθελα να σα παρέχω ω ανακοινώσει του Προέδρου. Τώρα θα προτείνω να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, αριθμό 3. Ανταλλαγή απόψεων με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή της Frontex σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση με τις γειτονικέ χώρες και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλάμε για μετανάστες και πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, ειδικότερα στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωση, καθώς και στο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεδομένων των συμβαντών της, Αραβική της Αραβικής ε, Άνοιξης και όλων των γεγονότων γύρω από τη Μεσόγειο. Παρακολουθούμε όλα αυτά τα συμβάντα καθώς και το τι συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά σύνορα ο κύριος καθηγητής Μπέντερ πέρυσι ε, διεξήγαγε μια μελέτη όσον αφορά τις επιπτώσεις των μεταναστευτικών πολιτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Γειτονία. Παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2011 σε εμάς, θα θυμάστε, ότι οδήγησε σε μια ε, αρκετά ζωηρή συζήτηση. Σύμφωνα με τη μελέτη υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για το, κατά πώς, ε, διαχειρίζεται τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σίγουρα κάποιες θετικές επιπτώσεις ε, στις εθνικές ε, προσεγγίσεις της διαχείρισης της μετανάστευσης. Ωστόσο υπάρχουν πολλά αρνητικά γεγονότα όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών. Παρότι όλες οι χώρες ε, στην ευρωπαϊκή γειτονία και οι υποένταξη χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο στην ανάπτυξη των μεταναστευτικών πολιτικών, τόσο στο πλαίσιο της νόμιμης όσο και της παράνομης μετανάστευσης. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ε, ακόμη θεωρούνται μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες, διότι τα ε, ανθρώπινα δικαιώματά τους παραβιάζονται τακτικά. Αυτοί οι άνθρωποι, οι μετανάστες, δεν έχουν καμία δυνατότητα να απαιτήσουν τήρηση των δικαιωμάτων τους και να αναζητήσουν νομική προστασία. Ακούμε από διάφορες πηγές πληροφορίες για το πώς ε, ε, ε, πραγματοποιείται κατάχρηση των δικαιωμάτων των μεταναστών. Τα βλέπουμε στις οθόνες των τηλεοράσεών μας σχεδόν καθημερινά. Στο φάκελο της συνεδρίασης θα βρείτε μια σύνοψη της μελέτης που σας ανέφερα μαζί με μια λίστα συστάσεων στο πλαίσιο της διμερούς οικονομικής συνεργασίας και ορισμένες πρακτικές πτυχές όλων αυτών η συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών μετανάστευσης ε, αποτελεί ζήτημα ανησυχία και θέτει ορισμένα ερωτήματα και κάποιες αμφιβολίες. Πρέπει να αναφερθεί ότι πριν από ένα σχεδόν χρόνο παρουσιάσαμε μια γνωμοδότηση στην ΑΦΕΞ για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Πρόκειται για, για μια γνωμοδότηση σε σχέση με τον νέο κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex που αφορούσε λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση ακριβώς αυτό το θέμα τη συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών μετανάστευσης. Σε αυτή τη γνωμοδότηση η διευρυμένη εξωτερική εντολή της Frontex αποτελεί θέμα ανησυχίας από όψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτή τη γνωμοδότηση καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Frontex και τρίτων χωρών. Σήμερα έχουμε εξέχοντες προσκεκλημένους κατά τη συνεδρίασή μας, όπως ανέφερα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερμά θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Φρανσουά Κρεπό που είναι ο ειδικό εισήγητη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Οι μας αυτή τη στιγμή, ο καλεσμένος μας αυτή τη στιγμή ασχολείται με τη μεσογειακή πτυχή του όλου ζητήματος στο έργο του και προσπαθεί να απαντήσει ερωτήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια έκθεση που αυτός θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών τον Ιούλιο του 2013. Καλώς ορίσατε λοιπόν και πάλι. Είμαι βέβαιος ότι θα μιλήσετε για τους στόχους και το πεδίο του έργου σας καθώς και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική στον χώρο της Μεσογείου. Οι προκλήσεις αυτές ε, προκαλούν δέος, ειδικότερα μετά από την Αραβική Άνοιξη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο, τον κύριο Γκέλ Άρες Φερνάνδες ε, αλλά αναπληρωτή διευθυντή της Frontex που δέχτηκε την προσκλήση μα ο κύριος Άρια. θα μας παρουσιάσει τι τελευταίες εξελίξει στη Frontex ειδικότερα ε, σε σχέση με τα καθήκοντά του αλλά και σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών. Κατά τη συζήτηση θα δώσουμε επίσης ε, το λόγο στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενημερώθηκα ο κ. Ντάριντε Τέμεμαν από την Γενική Διευθύνση Ιστορικών Υποθέσεων είναι παρόν. Θα έχετε λοιπόν... Θα βομβαρδιστείτε λοιπόν με ερωτήσεις και θα λάβετε το λόγο εν ευθέτω χρόνο. Χωρίς λοιπόν περισσότερη καθυστέρηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κρεπό ειδικό εισηγητή και αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των μεταναστών. Σας δίνω το λόγο. Και επίσης θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι έχουμε κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Παρακαλώ λοιπόν να περιορίσετε την ομιλία σας σε 8 λεπτά. Θα σας εμείνει ιδιαίτερα ευγνώμη. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και θα ήθελα να σας παρουσιάσω καταρχάς το έργο μου και μετά την αποστολή να σας παρουσιάσω ποιες θεωρώ ότι είναι οι προκλήσεις ε, στο κίνημα αυτό της αποστολής. Καταρχάς, ο ειδικός εισηγητής είναι εμπειρογνώμονας ε, που διορίζεται για τριετή περίοδο έχω καθολική εντολή για να ερευνήσω και να διερευνήσω θέματα μεταναστών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, να σας πω ότι αυτά είναι τα βασικά μου καθήκοντα και ασφαλώς είμαι υπεύθυνος και για άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά για θέματα επικοινωνίας, αποστολή επιστολών σε ε, διάφορες χώρες, έρευνες ε, για νομοθεσίες και το καθεξής. Με υποστηρίζει ο ειδησικός, ε, μάλλον το γραφείο του εισηγητή για το ΟΗΕ και η αποστολή μου έγκυται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είχα μία αποστολή το Δεκέμβριο στην Αλβανία, όπου διαπίστωσα τις συνέπειες της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα αυτή. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία. Και φέτος, μετά από την εμπειρία λοιπόν αυτή, αλλά και την προηγούμενη μου έρευνα που είχα διεξάγει, αποφάσισα να διερευνήσω το θέμα των ε, συνόρων τη Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα παγκόσμιο ε, φορέα, ε, το φάρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές προς την ε, περιοχή. Είναι πιο έντονη η πολιτική εστίαση στην περιοχή και έχουμε δυστυχώς και όλο και πιο πολλές αναφορές για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισκέπτομαι αυτή την εβδομάδα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, πήγα στη Βιέννη την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε λάβει ε, άδεια να μεταβούμε στην Τινησία τον Ιούνιο. Αναμένουμε απαντήσεις από την Τουρκία, επίσης για τον Ιούνιο και θα μεταβώ επίσης στην Ιταλία το φθινόπωρο και ελπίζουμε να μεταβούμε και στην Ελλάδα. Περιμένουμε απάντηση ε, το φθινόπωρο για να ερευνήσουμε το θέμα της Τινησίας και της Ιταλίας, των συνόρων και της Ελλάδας και της Τουρκίας ως ε, παράδειγμα για τα ευρωπαϊκά σύνορα θα υποβάλω αναφορά στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Ιούνιο και επίσης ε, θα έρθω και στι Βρυξέλλες να υποβάλω σχετική αναφορά. Λαμβάνουμε τακτικές εκθέσεις για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών που προσεγγίζουν, διασχίζουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες ε, ακραίες περιπτώσεις ε, περιλαμβάνουν θάνατο μεταναστών στην Μεσόγειο, για παράδειγμα, στην διαδικασία που διασχίζει τα σύνορα. Έχουμε φυσικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από συνοριοφύλακες. Αυτό δεν είναι τεράστιο ζήτημα ουσιαστικά, αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ε, μεγάλες περιόδους κράτησης, κράτηση υπό μη ανθρώπινες συνθήκες, ανηλίκων και το καθεξής. Αφενός, οι παραβιάσεις αυτές μπορεί να συμβούν σε επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γενικά είναι πιο εύκολο να παρακολουθηθούν, να δοθεί και να αποδοθούν ευθύνες ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που μας ενδιαφέρει όμως επίσης είναι τι συμβαίνει στα ίδια τα σύνορα και τι συμβαίνει και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συμβαίνει δηλαδή όταν προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα οι μετανάστες, για παράδειγμα στην Τουρκία και στην Τινησία. Θα τις ερευνήσουμε και τις δύο περιπτώσεις, γιατί και οι δύο χώρες ε, έχουν μεγάλες ροές τελευταία μεταναστών που προσπαθούν να εισάλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Τουρκία από την Ανατολή στην Τινησία από την υποσαχάρια Αφρική. Και θέλω να διερευνήσω λοιπόν πώς ε, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν, προωθούν, αποτρέπουν τις παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιώματων των μεταναστών. Αυτό λοιπόν μπορεί να συμβεί με διαφόρους τρόπους αυτή η επιρροή από πλευράς των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για παράδειγμα μέσω υποστήριξης ε, μέτρων που μπορεί να οδηγούν τα, κράτη, τα, κράτη να μην ε, καταγράφουν τέτοιες παραβιάσεις ή όταν υποστηρίζονται πολιτικές που δεν ε, βάζουν στο επίκεντρο τα δικαιώματα και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών. Υπάρχει φυσικά και θετικό αντίκτυπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υποστηρίζει η Ένωση, για παράδειγμα, με κυβερνητικές οργανώσεις, ε, ε, δικαστικές διαδικασίες και το καθεξής. Το θέμα είναι αυτό αποτελεί προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα βρεθεί ένα μοντέλο διαχείρισης των συνόρων, το οποίο θα συνάδει με μια προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και γίνεται μεγάλη εκταμένη αναφορά στα έγγραφα των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σύστημα παροχής ασύλου και την ενίσχυση αυτού του συστήματος σε όμορες χώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όντως να γίνεται και ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θετικός παράγοντας στην διαδικασία αυτή. Ωστόσο το άσυλο είναι ένα μικρό κλάσμα αποτελεί μάλλον και εκπροσωπεί ένα μικρό κλάσμα των μεταναστών που έρχονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επαρκεί να αντιμετωπίσουμε μόνο αυτές τις μεταναστευτικέ ροές. Δεν είναι η πλειονότητα. Οι πιο πολλοί είναι μετανάστες που δεν χρειάζονται τέτοιου είδους προστασία. Μπορεί να χρήζουν άλλου είδους προστασία, αλλά όχι αυτή οι μετανάστες στο διεθνές δίκαιο έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι μας εδώ στην αίθουσα, εκτός από το ε, δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε και το δικαίωμα του να εισέλθουν στην επικρέτεια. Όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα, δικαιώματα ισότητας, απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης και το καθεξής ισχύουν εξίσου στους μετα... και τους μετανάστες υπό το διεθνές δίκαιο. Και αυτό δεν θα πρέπει να το αμελούμε. Αποτελεί το σημείο κλειδί. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν εξίσου και για τους μετανάστες. Τα βασικά θέματα που θεωρώ ότι έχουν ανακύψει είναι τα εξής. Πολιτικές ε, επιστροφής. Αναφέραμε κάποιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι λόγοι κράτησης τώρα, οι αιτίες κράτησης. Η κράτηση θα πρέπει να είναι πάντα το μέτρο τη τελευταίας προσφυγής, όχι η πρώτη λύση που θα έρχεται στο μυαλό μα, Η διάρκεια της κράτησης Συνήθω είναι μακρές οι περίοδοι, μήνε, χρόνια. Όροι, συνθήκες κράτησης εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτηση παιδιών, πολύ συχνά φαινόμενα αυτά. Εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτηση οικογενειών πρόσβαση σε δικηγόρους, πρόσβαση σε δερμηνέα, πρόσβαση σε σωστά δικαστικά μέτρα. Όλα αυτά συχνά δεν παρέχονται στους μετανάστες. Πρόσβαση στο σχολείο, σε υγειονομική περίθαλψη για παιδιά και για γυναίκες, ε, σε τρόφιμα, σε κατάλημα, σε εργασία, σε τελική ανάλυση. Και όταν εργάζονται, προστατεύονται από το εργατικό δίκαιο πώς προστατεύονται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Οι προκλήσεις λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εγγύς μέλλον με μία προσέγγιση στα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών διασφαλίζοντας ότι θα αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα των μεταναστών σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις όμορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά πολιτικές συνεργασίες, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι όντως τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών είναι κάτι το οποίο γίνεται σεβαστό. Να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές μας δεν ε, διώχνουν το πρόβλημα στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και μετά να λέμε ότι άμα δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι δικό σας πρόβλημα, να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα δίνουν προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Και τώρα, 8 λεπτά για τον κύριο Γκίλ Άριας Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που προσκαλέσατε τη Frontex ε, να λάβει μέρος στην ε, σημερινή συνεδρίασή σας. Καλημέρα σε όλους. Μετά λοιπόν την πρόσκληση που απευθύνατε στην ε, Frontex, διάρθρωσα και εγώ την ομιλία μου σε τέσσερα κύρια τμήματα, εστιάζοντα βέβαια περισσότερο στα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρώτο θέμα θα είναι οι εξελίξει που είχαμε πριν ε, τον νέο κανονισμό για την Frontex που τέθηκε σε ισχύ ε, το 2011. Δεύτερο σκέλος θα είναι το πώς ε, εκτελούνται οι νέες δράσει που προβλέπονται για το 2012. Τρίτο σκέλος διμερή συνεργασία με φορείς που ειδικεύονται σε ζητήματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τέταρτον συνεργασία με τρίτες χώρες. Ξεκινώ λοιπόν με το πρώτο κεφάλαιο, ήτι θεμελιώδη δικαιώματα, μία από τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει στις δραστηριότητε της υπόψη η Frontex αφού ξεκίνησε το τέλος του 2005 τις δραστηριότητές της. Ωστόσο, η πιο ορατή δράση έλαβε χώρα το 2011 πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμό Frontex. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τη στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το σχετικό σχέδιο δράση. Το Μάρτιο του 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Frontex ενέκρινε τη στρατηγική τη υπηρεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχε συνταχθεί από μια επιτροπή την οποία πάρτιζαν εξωτερικοί εταίροι, όπω παραδείγματο χάρη ο, Οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλοι οργανισμοί, εκπρόσωποι της Κομισιόν και εκπρόσωποι των κρατών μελών. Βασίζεται στο γεγονός ότι η Frontex θεωρεί πως ο σεβασμός και η πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν συνιστώσεις αναπόσπαστα τμήματα μιας αποτελεσματικής διαχείρισης των συνόρων για μια πλήρη και δομένη υλοποίηση της ε, στρατηγικής συγγνώμη, ένα σχέδιο δράσης εγκρίθηκε από το ΔΣ της Frontex ε, το Σεπτέμβριο του 2011 και στο σχέδιο αυτό υπάρχουν 20 δράσεις με τις οποίες η Frontex θα υλοποιήσει την στρατηγική. Μεταξύ αυτών συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους. Οι δράσεις έχουν να κάνουν με τις βασικές δραστηριότητες ε, της Frontex, επιχειρησιακές δηλαδή, ε, ανάλυση κινδύνων, επιχειρήσεις, ε, δημιουργία υποδομών, αλλά και οριζόντιες δραστηριότητες. Εξωτερικές σχέσεις, ε, επικοινωνία κτλ. Δεύτερον, κώδικας διοντολογίας της Frontex. Η Frontex έχει εκπονήσει ένα κώδικα διοντολογίας που χρησιμοποιείται στις ε, δραστηριότητες τη επιχειρήση της και ισχύει για όλους όσους συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες της Frontex. Κατάρτιση, συναντήσεις και το καθεξής. Περιλαμβάνει επίσης και κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του κώδικα διοντολογίας. Μπορεί δηλαδή αυτό να σημάνει και άμεση απομάκρυνση εν λόγω ατόμου της δραστηριότητα ε, της Frontex. Επίσης η Frontex ε, εξετάζει και αναθεωρεί τον κώδικα δεοντολογίας αυτή τη στιγμή εν ώψη της υλοποίησης του νέου κανονισμού Frontex. Το 2α άρθρο του κανονισμού αναφέρεται στον κώδικα διοντολογίας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ε, ομάδων των ε, κοινών, ε, της κοινή στήριξη και της ε, ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Έχουμε ένα νέο όνομα πλέον, το οποίο καθιερώνεται με το νέο κανονισμό. Θα, υπάρχει, λοιπόν, θα υπάρχουν αυτές οι ομάδες με συνοριοφύλακες, εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης των συνόρων. Τα κράτη-μέλη θα συνεισφέρουν στην δεξαμενή, αν θέλετε αυτή, με βάση συγκεκριμένα προφίλ τα οποία εκπονεί Frontex μετά τον ορισμό και τη συμπερίληψή του σε αυτήν την ομάδα θα παρέχει Frontex κατάρτιση στα μέλη της ιδίως σε σχέση με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θεμελιώδη δικαιώματα, πρόσβαση στη διεθνή προστασία και το καθεξής. Το δεύτερο σκέλος παρουσίασής μου τώρα αφορά την υλοποίηση του τροποποιημένου το 2012 κανονισμού Frontex. Είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και ε, θα ξεκινήσω με τον ε, Human Rights ε, Officer. Στο άρθρο 26α, ο κανονισμός δίνει την εντολή στην Frontex να δημιουργήσει ένα συμβουλευτικό φόρουμ και να ορίσει έναν υπεύθυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, Fundamental Rights Officer. Το ε, Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν έχει συγκροτήσει μια συμβουλευτική επιτροπή την οποία απαρτίζουν εκπρόσωποι του ΔΣ από διάφορα κράτη-μέλη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εκπρόσωποι των ε, οργανώσεων εταίρων όπως ο Οργανισμός των Μιλτών Δικαιωμάτων, το Γραφείο Υποστήριξης ε, της, του Ασύλου και το UNHCR, η Πατέρα Μαστήλα της Καθοδηγείται λοιπόν ε, ο οργανισμός για την υλοποίηση του άρθρου αυτού που σας προανέφερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συμβουλευτικό φόρουμ, αυτό θα έχει ως αποστολή να βρεθώ τον εκτελεστικό διευθυντή και το ΔΣ σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα γνωμοδοτεί για περαιτέρω εξελίξεις και την ανάπτυξη και την υλοποίηση τη στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κώδικα δεοντολογίας. Προβλέπουμε δύο βασικά να είναι τα είδη των συμμετεχόντων, τύποι των συμμετεχόντων. Πρώτη ομάδα, οργανώσει κοινωνία των πολιτών. Θα είναι η πλειοψηφία. 9 στα 15 μέλη τη επιτροπή αυτή, του Φόρουμ, συγγνώμη. Δεύτερη ομάδα, διεθνείς οργανισμοί και οργανισμοί της Ένωσης που ειδικεύονται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τρεις ε, οργανισμοί υποχρεωτικοί, το αναφέρει δηλαδή συγκεκριμένο κανονισμός, ΕΑΣΟ, Οργανισμός ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, UNHCR και η Συντακτική Επιτροπή προτείνει τον IOM, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε μια απόφαση για τη σύνθεση του ε, συμβουλευτικού, μάλλον θα λάβει τη συμβουλευτική, την ε, πρόταση για το συμβουλευτικό φόρουμ ε, αυτό το μήνα, στις 12 συγκεκριμένα του μήνα. Επίσης θα υπάρξει και ένα ανεξάρτητο μέλος που θα είναι υπεύθυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα έχει ως καθήκον να αναφέρει τακτικά και, στην, και στο Συμβουλευτικό Φόρουμ τον υπεύθυνο αυτόν θα τον ορίσει το ΔΣ της Frontex, κάτι που αναμένουμε για το Σεπτέμβριο στη συνεδρία του ΔΣ. Είχε δημοσιευτεί η θέση και ο ή υποψήφιο θα αναλάβει τα καθήκοντά του της πριν τα τέλη του 2012. Ο υπεύθυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα θα έχει μία ε, έναν εποπτικό ρόλο. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω την πρόταση για τη διαδικασία λήξη ή αναστολή κάποιων επιχειρήσεων σε περίπτωση καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κανονισμό έχει μια ρήτρα για τακτική εξέταση των επιχειρήσεων για να δούμε κατά πόσο ε, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το άρθρο 3 ορίζει ότι ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού της Υπηρεσίας θα μπορεί να αναστείλει ή να ε, πάυσει κάποια πιλωτικά προγράμματα, είτε μερικά είτε εξ ολοκλήρου, εάν υπάρχουν ε, παραβιάσεις ε, των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Για να τηρήσει η Frontex αυτές τις διατάξεις, αυτή τη στιγμή ε, αναπτύσσει έναν εσωτερικό μηχανισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία και ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις φάσεις, από τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων μέχρι την ε, ολοκλήρωσή τους ή την πάυση τους. Σε ό,τι αφορά τη διμερή συνεργασία με άλλους εταίρους, άλλους οργανισμούς, η Frontex και η UNHCR, με τη UNHCR, την Πατρεμοσία για τους Πρόσφυγε, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία Έχουμε προετοιμάσει από κοινού ε, μια, ένα πρόγραμμα κατάρτισης ε, για τους ε, πρακτορές μας. Σε ό,τι αφορά τον οργασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, πιστεύω ότι είναι αμοιβαία επικοδομητική συνεργασία μας. Με την εμπειρογνωμοσύνη της μας βαθά ο οργανισμός αυτός να μεταφέρουμε στην πράξη ε, τη θεωρία στην σχετική με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ εμείς παρέχουμε στήριξη στο έργο του ΦΡΑ. Και επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη, στην κατάρτιση, σε κάποια εγχειρίδια βέλτιση των πρακτικών και επιχειρησιακό επαγγελματικό κώδικα διοντολογίας για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωματών. Ο ΦΡΑ βοήθησε επίσης και στη σύνταξη ε, του καταστατικού για τα, άνθρωπα, δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ΕΑΣΟ. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας το 2011. Η Frontex συμμετέχει και συνεισφέρει ε, στις ε, συνεδριάσεις του ΔΣ. Συνεδριάζουν κάποιες μονάδες ε, της Frontex με τους εμπειρογνώμονες του ΕΑΣΟ, όπως και φέτος έγινε αυτό, για να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε με στόχο να υπογράψουμε έναν διακανονισμό εργασίας Τέλος, συνεργασία με τρίτες χώρες. Πρωταρχικός στόχος της Frontex είναι η εντατικοποίηση της εφιστάμενης διμερού συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες και χώρες προέλευσης ή διέλευσης παράνομων ε, μεταναστών. Λαμβάνεται υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα ο χάρτης των δημιουργών δικαιωμάτων. Επίσης, συνεργαζόμαστε με υποψήφιες ή δυνητικά υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στόχος μας μεταξύ άλλων είναι να έχουμε μια καλή ε, διάρθρωση της ε, διαχείρισης των συνόρων σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και έχουμε την ε, διέλευση δια της θαλάσσης και η Μεσόγειος είναι πάρα πολύ στο επίκεντρο όλων αυτών των προσπαθειών της Frontex. Έχουμε ξεκινήσει σχέση με 16 χώρες, διαπραγματεύσεις επίσης με αρχές ακόμη 9 χώρων έχουμε ξεκινήσει και έτσι ολοκληρώνω την παρέμβασή μου κύριε Πρόεδρε και βεβαίως με θυμάσαι να στα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Άρια και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να ξεκινήσει η συζήτηση. Η κυρία Λόχ Μπίλερ, η πρόεδρος της Επιτροπής μας, θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ και συγγνώμη που καθυστέρησα. Άκουσα όμως τις παρουσιάσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και συγκεκριμένα προς τον κύριο Κρεπό, αλλά και για τον κύριο Φερνάντες. Κάποιες φορές ε, και στη δική μου χώρα, τη Γερμανία, υπάρχει κάποια πολιτική ε, διάθεση να προστατευτούν οι μετανάστες, ε, να προστατευτούν από ενδεχόμενο κίνδυνο, να δημιουργηθεί ένα κέντρο υποδοχής, όπως αποκαλείται, προκειμένου να, να καταφέρουν να έχουν τέτοια δικαιώματα από πλευρά ε, του Μαγκρέμπ. Είσαστε υπέρ μια τέτοια ιδέα. Γιατί το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα διακινδυνεύουν ε, τη ζωή τους ε, χρησιμοποιώντας μια εγκληματική οργάνωση. Κατά δεύτερον, μας είπατε ποιες χώρες θα επισκεφτείτε και είναι σαφές ότι η κατάσταση είναι αρκετά δραματική σε αυτές. Να σας ρωτήσω όμως, παρακολουθείτε όμως και την κατάσταση στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα σύνορα στην Ουκρανία. Κανένα από τα κρατημέλη μας δεν έχει επικυρώσει την ε, συνθήκη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των μεταναστών και για τις οικογένειές τους. Είναι κάτι σημαντικό, αυτό θεωρείτε. Και ένα ερώτημα και προς τους δύο ομιλητές. Ακούσαμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά μια υπόθεση κατά της Ιταλίας. Ακούσαμε ότι κανένα μέρος στον κόσμο δεν αποτελεί τοποθεσία όπου δεν δίνεται σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας βοηθάει αυτή η απόφαση γιατί όταν καταρτήσαμε τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον της Frontex, πάντα αυτό το νομικό ζήτημα του ποιου δικαίου ισχύει δεν ε, κατάφερνε να επιληθεί. Τώρα θεωρώ ότι έχει γίνει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό επηρεάζει το έργο σας και για σας κυρία Αρίας. Είπατε ότι από το 2005 που ξεκίνησε το έργο της Frontex θεωρείτε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικό τμήμα της δουλειάς σας. Πάρα πολύ ε, θετικό αυτό, γιατί νομίζω ότι ένας προηγούμενος ε, γενικός διευθυντής της Frontex ε, είχε δηλώσει σε επίσκεψη στο Κοινοβούλιο ότι δεν έχει η Frontex αρμοδιότητα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα λοιπόν έχετε μια καινούργια εντολή. Αν προκύψουν υποθέσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από προσωπικό της Frontex. Πώς πρόκειται να το αντιμετωπίσετε, γιατί πλέον έχετε κώδικα την εντολογίας, μας είπατε. Αυτό ίσχυε και πριν το 2011 και ένα σχόλιο, επιτρέψτε μου, δεν με ικανοποιεί να λέτε ότι Ίσως μέχρι το τέλος του 2012 να καλύψετε τη θέση του αρμόδιου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι κατεπήγον, θεωρούμε. Ακόμα και η ίδια η θέση είναι αμφιλεγόμενη, γιατί θα θέλαμε έναν ανεξάρτητο τέτοιο αρμόδιο, ενώ η θέση αυτή που έχει προκριχθεί ουσιαστικά θα πρέπει να περιέχει κάποιον ο οποίος θα υποβάλει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ την Πρόεδρο. Η κυρία Κέλλερ ζήτησε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ερωτήσεις και προς τους δύο σας. Ε, κύριε Κρεπό, δεν γνωρίζω αν έχετε ακούσει για τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη δημιουργία του Eurosur, ε, Ευρωπαϊκό Εποπτικό Σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα συνιστώσεις ε, όπως συντονισμό εντός των κρατών μελών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπλέον διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, ειδικότερα με την Τινησία, τη Λιβύα και ούτω καθεξής γύρω από τη Μεσόγειο και κυρίως στο νότιο της μέρος και επίσης περιλαμβάνει μια συνειστόσα επιτήρηση των συναριακών περιοχών, ειδικότερα της Μεσογείου με μεγάλες ποσότητες τεχνικού εξοπλισμού. Έτσι λοιπόν η Frontex και τα κράτη-μέλη όταν θα αντιλαμβάνονται ε, ύποπτες αναχωρήσεις ε, σκαφών από την Τινησία μπορούν να ε, ενημερώνουν τις ακτοφυλακές της Τινησίας και να τους ζητούν να σταματούν αυτά τα σκάφη. Έτσι λοιπόν μπορεί να παραβιάζονται το δικαίωμα αναχώρησης από μια χώρα καθώς και μπορεί να παραβιάζεται η ε, οδηγία μη επιστροφής. Ε, πώς θα είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι δεν θα παρεμβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτό το πλαίσιο. Και όσον προς τον κύριο Άρια Φερνάνδε, ε, ε, κάνω τι ίδιε ερωτήσει με την κυρία Λοχπίλερ για ποιο λόγο πήρε τόσο πολύ καιρό και ακόμη δεν έχουμε επιτύχει ακόμα να έχουμε ένα απλό αξιωματούχο Ευρωπαίο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρχε στο σχέδιο ε, ανέκαθεν, το έχει περάσει πάνω από χρόνος και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει θα ήθελα να πείτε γιατί έχει πάρει τόσο πολύ καιρό το ίδιο και για το Συμβούλιο. Ε, είναι τόσο δύσκολο να δημιουργήσετε μια δομή που θα σας πάρει συμβουλευτική υποστήριξη. Επίσης είπατε ότι μελετάτε ένα σχέδιο κριτηρίων για τις συνθήκες ε, αναστολής ή τερματισμού δραστηριότητας ε, όταν πληρούνται κάποια κριτήρια. Έχουμε ακούσει τα ίδια από τον κύριο Λάιτινεν πριν από πολλούς μήνες στην Επιτροπή Λίμπε όπως φαίνεται λοιπόν η διαδικασία όλη αυτή έχει διαρκέσει ήδη έξι μήνες και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει. Και τι κάνετε σε σχέση με τις τρέψεις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακούσαμε όλοι για το τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά σύνορα, τις σχετικές παραβιάσεις, οι οποίες είναι πολύ καλά τεκμηριωμένες, αλλά αντί να σταματήσουμε τις δραστηριότητες της Frontex εκεί, απλά αξιολογείται τα κριτήρια αλλά δεν πάβουν να γίνονται παραβιάσεις ε, συνεχώς ε, σε αυτή την περιοχή απαράδεκτη είδου. Για ποιο λόγο λοιπόν το αφήνετε να συνεχίσετε και τι κάνετε με όλες αυτές τις περιπτώσεις παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχετε κάποιο σχέδιο κριτηρίων, έχετε την πραγματικότητα μπροστά, τας, μπροστά σας και ακόμη μιλάτε θεωρητικά. Πώς ε, γίνονται λοιπόν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιο άλλο να λάβει το λόγο. Υπάρχουν ερωτήσει. Έχω εγώ μία ερώτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σχετική, αλλά ακούγοντας ε, και τους δύο μιλητές αναρωτήθηκα κατά πόσο αντιπροσωπεύεται δύο αντίθετα μέρη από τη φύση τους. Όταν ακούω να μιλάνε για τη Frontex και τις δραστηριότητες της, ε, στο μυαλό μου έρχεται ε, ένας οργανισμός ε, πρόληψης και καταστολής μάλιστα που ουσιαστικά προστατεύει το φρούριο της Ευρώπης ε, από τους ανθρώπους που έρχονται και που αν δεν τους σταματήσουμε ε, ότι και τους οποίους μπορούμε να σταματήσουμε μόνο με μέτρα καταστολής και αστυνόμευση ακούγοντάς σας κύριε Κρέπο χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα ότι επιμένετε ακόμη ότι οι μετανάστες έχουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα και λοιπά δικαιώματα όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι αλλά ε, κοιτώντας ε, τους χώρους συγκέντρωσης, ε, τους χώρους διαμονής τους, τις διάφορες πρακτικές ε, ε, αντιλαμβανόμαστε ότι ισχύει το, ακριβώς το αντίθετο από όσα λέτε όσον αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστών οι οποίοι βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση όπως φαίνεται μάλιστα η κατάστασή τους γίνεται όλο και πιο απελπιστική. Αναρωτιέμαι πώς εσείς ε, θεωρείτε τις δυο σας απόψεις και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ήταν πολύ ενδιαφέρον που βρίσκεστε και οι δύο μαζί ταυτόχρονα σε αυτή την Επιτροπή. Συνεργάζεστε μαζί και προσπαθείτε να εναρμονίσετε αυτές τις δύο προσεγγίσεις ε, όσον αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και την κατάστασή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να κάνει κάποια ερώτηση. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι επίσης ε, επικροτώ το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία συνεδρίαση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, ε, από τη μία πλευρά, Έχουμε αντιπροσώπους ενός οργανισμών που ασχολούνται με τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και από την άλλη πλευρά έχουμε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό αρμόδιο για την τήρηση και το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων. Αυτή η κατάσταση ήρθε στο φως μετά από την Αραβική Άνοιξη, μετά από την οποία αυξήθηκε η μεταναστευτική πίεση τόσο από τις χώρες ε, όπου έλαβε χώρα η Αραβική Άνοιξη στη Βόρεια Αφρική, όσο και από άλλες χώρες. Και άλλοι μετανάστες εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία, την κατάσταση, για να προσπαθήσουν να ε, μεταναστεύσουν στην Ευρώπη. Άνθρωποι από χώρε με περίπλοκη και χαοτική εσωτερική κατάσταση, οι άνθρωποι που μεταναστεύουν στην Ευρώπη από τη Λιβύη, για παράδειγμα, ε, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση τραυματικές εμπειρίες εδώ λοιπόν ε, δεν έχουμε απόλυτα σωστή εικόνα της κατάστασης. Έχουμε ακούσει πολλά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, μιλάμε όμως για πολύ ε, για προγράμματα που προβάλλονται αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί διότι δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή ωστόσο δείχνουν την κατάσταση των μεταναστών σε χώρες όπως η Ελλάδα για παράδειγμα. Ε, όλο αυτό συνοδεύεται από μια δυσχερή οικονομική κατάσταση που επίσης ε, ε, παρεμποδίζει και περιορίζει τις δυνατότητες αυτών των παραμεθοριών, των παραμεθοριών χωρών. Σχετίζεται αυτό με τα προβλήματα χρηματοδότησης κέντρων για πρόσφυγες και μετανάστες. Όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, για πολίτες γειτονικών και χωρών και χωρών της Νοτιού Μεσογείου είναι πολύ σημαντική, ειδικότερα μετά από την υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονό ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης καθιερώθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα θεσμικά όργανα να συντάξουν ένα σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Κομισιόν ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση αυτού του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά. Το σχέδιο δράσης αυτό δεν είναι πανάκια και δεν θα επιλύσει απαραίτητα όλα τα ζητήματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματο. Θα ήθελα λοιπόν να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να ρωτήσω τον κύριο Αρία Φερνάνδε ε, για το ακολουθό ζήτημα. Από δική μου εμπειρία γνωρίζω ως ε, πρόεδρος ε, της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην Πολωνία. Η εμπειρία μου δείχνει ότι η Frontex ε, δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με τα εθνικά κοινοβούλια. Τουλάχιστον τρεις φορές ε, καλέσαμε τον διευθυντή της Frontex ε, να παρευρεθεί στο κοινοβούλιο και τις τρεις φορές δεν τα καταφέραμε. Θα έλεγα ότι αυτή η συνεργασία μεταξύ του οργανισμού Frontex και των κρατών μελών ειδικότερα με τις Επιτροπές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εσωτερικών Υποθέσεων Χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν θα είναι δυνατόν να διεξαχθεί αυτός ο διάλογος. Από όσα είπε ο κύριος Άρες Φερνάντες, φαίνεται ότι έχετε αναλαβεί πολλές δεσμεύσεις ε, σε σχέση με την αύξηση και τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Όπως υπόθηκε, η μεταναστευτική πίεση αυξάνεται. Έτσι θα ακολουθήσουν όλο και περισσότερα προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού αυτού, της Frontex, του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν αλλά και με τα εθνικά κοινοβούλια στα κράτη-μέλη μια, τόσο, μια καλή συνεργασία θα παρήχε την απαραίτητη προστιθέμενη αξία. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να επισημάνω το πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία. Πιστεύω ότι οι ιδέες και οι έννοιε που παρουσιαστεί εδώ παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα συμβάλλουν σε καλύτερα πρότυπα, σε καλύτερη αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και κάποιοι αντικειμενικοί παράγοντες, ε, για παράδειγμα εκλογές. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι υπάρχει αρνητική στάση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους μετανάστες. Ίσως να μην μιλάμε απλά για έλλειψη φιλοξενίας, αλλά ουσιαστικά για εχθρότητα. Όταν υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα, συχνά αντιμετωπίζουμε ως αποδιοπομπαίο τράγο, τράγο τους ανεπιθυμητούς καλεσμένους μας και αυτό ισχύει ειδικότερα για μετανάστες σε χώρες ε, όπου, οι οποίες πλήττονται από διενέξεις. Αυτό είναι αναπόφευκτο, είναι μια δύσκολη ε, κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η δική μας Επιτροπή έχει ιδιαίτερη ευθύνη από αυτή την άψη και όπως είπε ο κ. Σκάρα και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αντιμετωπίζει επίση τη μετανάστευση ως ε, ζήτημα θεμελιώδου σημασία διότι οι μετανάστες όταν συλλαμβάνονται ε, και ε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται σχετίζεται με τις εσωτερικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Τόμπι Κίνγκ ε, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Προτείνουμε τρία λεπτά, εάν σας αρκούν. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω λίγο για τον τρόπο με τον οποίο η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή θα μιλήσει για τα θέματα της Frontex. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την εξής ε, θέση σε ό,τι αφορά την εξωτερική δράση στον ε, κλάδο της ελευθερίας δικαιοσύνης ε, σε ό,τι αφορά τις μονοταλιστικές ροές, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει βασική θέση. Και είναι σημαντικό αυτές οι χώρες στην διαδικασία κατάρτισης των σχέσεων να σέβονται τα δικαιώματα αυτά σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης ε, θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ολιστική και συνολική η προσέγγιση μας για να διασφαλίσουμε σε σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, σε πρόσφατη ανακοίνωση του Νοεμβρίου του 2011 για την καθολική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κινητικότητα τη μεταναστευτική που ορίζει το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η ανακοίνωση λοιπόν τονίζει πόσο σημαντικό είναι να τίθεται στο επίκεντρο ο μετανάστης ε, στο επίκεντρο της ανάλυσης γιατί το θέμα δεν είναι οι ροές, είναι ο άνθρωπος. Οι μεταναστευτικές ε, πολιτικές λοιπόν θα πρέπει να αποκρίνονται στις φιλοδοξίες και στις ανάγκες του κόσμου τον οποίο αφορούν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια καθολική προσέγγιση, να ενισχυθούν τα δικαιώματα των μεταναστών στις χώρες από που προέρχονται, στις χώρες προορισμού και στις χώρες τις οποίες διασχίζουν. Θα πρέπει λοιπόν ο διάλογος να προσπαθήσει να διασφαλίζει τα δικαιώματα αυτά σε όλη τη διαδικασία της μετανάστευσης. Επίσης, η ανακοίνωση υπογραμμίζει δύο βασικά προβλήματα, δύο ιδιαίτερα προβλήματα για πρώτη φορά να γνωρίζετε η σημασία των ανθρώπων που δεν έχουν πατρίδα. Και επίσης ε, θα πρέπει να τονιστεί και το θέμα το, της παράνομης κράτησης των μεταναστών σε τρίτες χώρες. Συνεργαζόμαστε λοιπόν ε, με τις άλλες υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Στις επαφές μας με τις τρίτες χώρες για τα δικαιώματα των μεταναστών υπάρχουν δύο βασικοί οδοί διαλόγου που χρησιμοποιούνται υπό επιτρεπές ε, για ιστορικά ζητήματα και για κοινωνική μετανάστευση που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής και για τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αποτελούν δική μας αρμοδιότητα. Και φυσικά τα δικαιώματα των μεταναστών προκύπτουν και στις δύο περιπτώσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν του διαλόγου αυτού στα σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αντιμετωπίζουμε θέματα όπως η συμπεριφορά των συνεργοφυλάκων. θέματα σε ό,τι αφορά την κράτηση των μεταναστών, τη βάση κράτησης, την ανάγκη να αποφευχθεί αυθαίρετη η κράτηση, η όρη κράτησης και σε ό,τι αφορά η πρόσβαση σε ενδικά μέσα σε ό,τι αφορά επίσης έχουμε θέσει το θέμα των ε, εργαζόμενων μεταναστών σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στον τομέα των οικοδομών και της ε, οικιακής ε, παροχής βοήθειας. Επίσης έχουμε θέσει και θέματα ασύλου όπου χρειάστηκε. Ένα παράδειγμα να σας δώσω για τα θέματα τα οποία θίγουμε με τρίτες χώρες, στις επαφές με τρίτες χώρες. Το Μάρτιο του 2003 του 2012 θέσαμε ένα ζήτημα για το Λίβανο, μια δήλωση μετά τον τραγικό θάνατο ε, Αιθιοπιού εργαζόμενου. Στην ε, δήλωση αυτή ε, εκφράσαμε τη λύπη για τη θάνατο της κυρίας αυτής και δώσαμε αρμοδιότητα πλήρους ε, έρευνας των αιτιών που οδήγησαν στο θάνατο της κυρίας. Τονίσαμε ότι χρειάζεται μηχανισμός προστασίας και νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο Λίβανο, προκειμένου να υπάρχει σωστή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να, να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματά τους. Και θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα, τα, τα ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης ε, των εργαζομένων αυτών. Αυτό αποτελεί ένα απλό παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να καλέσω τον κύριο Τέμερμαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Thank you, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι το τον συντομότερος. Είδαμε το 2011 κάποιες μεγάλες αλλαγές, όχι μόνο στις πολιτικές ε, τις οποίες έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και ε, στην κατανομή των αρμοδιοτήτων, όπως είπε και ο συνάδελφος ε, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η συνολική προσέγγιση των θεμάτων αυτών είναι σημείο κλειδί η προσέγγιση λοιπόν αυτή συνενώνει τις ε, συνέργειες των εμπειριών που ήδη έχει αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πρακτική στο εσωτερικό των κρατών μελών. Προσπαθούμε επίσης να προωθούμε μέσω ανακοινώσεων τις βέλτιστες πρακτικές σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις με τρίτες χώρες. Το 2011 ήταν επίσης το έτος κατά το οποίο είδαμε την υιοθέτηση του τροποποιημένου κανονισμού της Frontex. Και πρέπει να πω ότι από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούμε να πούμε ότι έγιναν και πάρα πολλά από την αρχή της έναρξης, αν θέλετε, της δραστηριότητες της Frontex το 2005, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι εργάζεται σε κενό νομικό η Frontex, γιατί θεωρούμε ότι πάντα υπόκειτο στην πλήρη προστασία των θεμελιδών δικαιωμάτων κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Δυστυχώς θα πρέπει να πω, και αυτό το τονίζουμε σε κάθε περίσταση, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, εθνικής αρμοδιότητας. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα και καθορίζουν την είσοδο στην επικράτειά τους. Η Frontex αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως σκοπό να διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά θέματα εξωτερικών συνόρων. Υπάρχει λοιπόν μία διαφορά στο σημείο αυτό, γιατί κάποιο είπε κατά τη διάρκεια τη συζήτηση ότι η, η Frontex είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων τη ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ, ακόμα και με το τροποποιημένο νομικό πλαίσιο, αυτό δεν ισχύει. Άρα, Αυτό το σημειώνω. Έχει γίνει πολλή δουλειά στον τομέα αυτό, αλλά πολλά απομένουν ακόμα να γίνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καθεαυτή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομίζω ότι πλέον είναι σαφές ότι πολλά θα πρέπει να γίνουν και εντός της Frontex η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ε, τους στόχους και τον απότερο σκοπό του να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία και να ε, πληρωθεί η θέση του υπεύθυνου για ανθρώπινα δικαιώματα και του Συμβουλευτικού Φόρουμ. Να σας ενημερώσω τώρα για το έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά την Eurosur. Πρόκειται για μια νομοθετική πρόταση η οποία βρίσκεται σε φάση συζήτησης στο Συμβούλιο. Νομίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εισέλθει και σε διαδικασία συναπόφασης και νομίζω ότι και στο σημείο αυτό βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, γιατί η εποπτεία των εξωτερικών συνόρων είναι κάτι που καλύπτεται ήδη από την φυστάμενη νομοθεσία. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε συνέργειες, αν θέλετε, όταν τα σκάφη που πλέουν στην Μεσόγειο μέσω συνεργασίας ε, κρατών μελών με αρμόδιες αρχές περί χωρών ε, θα μπορούν να αντισωθούν με περισσότερους τρόπους, με καλύτερο τρόπο, γιατί σε, στις περισσότερες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται κατηγορίες ότι η Frontex δεν καταβάλει επαρκείς προσπάθειες να σώσει τον κόσμο που προσπαθεί να τη διασχίσει την Μεσόγειο, η οποία μπορεί να είναι και πολύ δύσκολη, όπως ξέρετε. Αυτά λοιπόν είναι τα σχέδια και η παρουσίαση του που βρισκόμαστε σήμερα. Για το ερώτημα που θέσατε, Πρόεδρε, για το τι έχει γίνει ως τώρα, σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης, θα πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ΣΟΚΟΜ, έχει σημειωθεί κάποια πρόβλημα. Το πρόγραμμα της Στοκόλμης ε, υπάρχει κάποια πρόοδος και το σχέδια δράσης για τη μετανάστευση αποτυπώνονται πλέον όλες οι δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα αυτό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ασφαλώς τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν βασικό ζήτημα στο πλαίσιο αυτό. Ελπίζω να σας παρουσίασα λίγο πολύ λοιπόν όλα τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω τώρα να ζητήσω από τους προσκεκλημένους μας να απαντήσουν στα ερωτήματα και στα σχόλια. Ιδίως ό,τι αφορά κάποιες ε, κρίσεις, κάποιες αξιολογήσεις. Παρακαλώ, κύριε Κρέπο, έχετε πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω ανάποδα στα ερωτήματα, από το τέλος προς την αρχή. Κάποιος με ρώτησε αν είμαστε ε, αντιμέτωποι ένας προς τον άλλον ως φορείς. Όχι, στο ε, διεθνές δίκαιο υπάρχει ιδίω η εδαφική κυριαρχία, υπάρχει ανεξαρτησία των κρατών. Αυτό είναι κατοχυρωμένο και εμεί προσθέτουμε ένα παράδειγμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο παράδειγμα ε, του διεθνούς δικαίου. Από κοινού λοιπόν, χέρι με χέρι, η εθνική κυριαρχία με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παραδείγματα του διεθνούς δικαίου και θα πρέπει να μπορέσουν να συνεργαστούν και να ε, συμβιώσουν. Δεν είμαστε αντίθετοι ένα προς τον άλλον, μπορεί να είναι διαφορετικοί οι στόχοι μας, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε. Και όταν ε, λέω ότι, δεν περι... ότι μάλλον δεν θα πρέπει να περιορίζουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα την εδαφική κυριαρχία ούτε και το αντίστροφο. Είναι δύσκολη η εξέβρεση της ισορροπίας, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Για το Eurosur με ικανοποίησε αυτό που άκουσα. Βέβαια είναι λίγο μυστήριο για μένα. Δεν έχω αρκετές λεπτομέρειες. Ε, φαντάζομαι ότι είναι η αρχή αυτής της ε, επιχείρησης και θα ήθελα να μάθω περισσότερα. Θεωρώ ότι το Eurosur είναι ένα εργαλείο και θα πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιείται το εργαλείο αυτό. Περιμένω τα δικαστήρια κάποια στιγμή να κληθούν να κρίνουν κατά πόσον χρησιμοποιείται με σοφία και σύνεση το εργαλείο αυτό. Και θα πρέπει να υπάρξει εποπτεία. Έχουμε και εμείς τις δικές μας σκέψεις, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε πώς χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο και ε, εν συνεχεία να κρίνουμε. Και φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα βοηθήσουν ε, πάρα πολύ και τα δικαστήρια. Με χαρά επίσης άκουσα την πρόοδο που υπάρχει για αυτό το μηχανισμό για την εξωτερική πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, μετά το πρόγραμμα της Στοκόλμης δεν το είχα ξανακούσει. Χαίρομαι λοιπόν που γίνονται κάποια πράγματα και στο μέτωπο αυτό. Απόφαση Χέρση ανέφερε τα σχετικά κυρία Λόχμπιλερ. Πράγματι ισχύει ε, παντού. Υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και όπου ασκείται εξουσία ε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. Ε, ανθρώπινα δικαιώματα πηγαίνουν μαζί με την άσκηση της εξουσίας και εκεί ε, είναι και ο δικός μας ρόλος να τηρούνται πάντοτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οικονομικών μεταναστών και των οικογενειών τους. Είμαι πάρα πολύ ε, απογοητευμένος ε, προσωπικά. Νομίζω ότι στον ΟΗΕ ισχύει το ίδιο για το ότι οι χώρες συνολικά του Βορρά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση αυτή ακόμη. Το μόνο που κάνει ουσιαστικά ή λίγο παραπάνω είναι να επαναλαμβάνει αυτή η σύμβαση αυτό που ισχύει στο διεθνές δίκαιο. Και το εφαρμόζει στους μετανάστες. Όπως η σύμβαση για τα άτομα με αναπηρία. Ουσιαστικά προσπαθεί να επεξεργαστεί λίγο περισσότερο ε, τη λογική των όσων ήδη περιέχονται στι διατάξει του διεθνού δικαίου και να εφαρμόσει τι σχετικέ διατάξει στα άτομα με αναπηρία. Κάποιε φήμε φήμες ότι ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαν επικυρώσει αν δεν είχαν πάρει τηλεφωνήματα από άλλε πρωτεύουσε, Είναι κάτι που ακούγεται, δεν ξέρω κατά πόσο αναλυθεύει η φήμη αυτή. σω οι χώρε οι σχετικέ θα μπορούσαν να το επιβεβαιώσουν να το διαψεύσουν. Εγώ πάντως θα ήθελα να ενθαρρύνω όλα τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν αυτή τη σύμβαση. Γιατί η σύμβαση αυτή σημαίνει, και αυτό σημαίνει και κύρωση αυτή τη σύμβαση. σημαίνει ότι υπάρχει ουσιαστική και σοβαρή δέσμευση όλων για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μεταναστών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επαναλαμβάνω. Όλοι οι μετανάστε έχουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα και αυτοί που δεν έχουν επίσημα έγγραφα. Έχουμε το κεφάλαιο 4, αν δεν απατώμε, τη σύμβαση που αναφέρει τα δικαιώματα όλων των μεταναστών και το κεφάλαιο 5 μιλά για κάποια επικουρικά, κάποια συμπληρωματικά δικαιώματα για μετανάστες που βρίσκονται, ε, που είναι νόμοι. Άρα τι θα πει αυτό, ότι το 4 ισχύει και για του μη νομίμω Αυτό είναι ο σκόπελο. Εκεί κολλάνε τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν να επικυρώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, σύμβαση αυτή. Εμεί όμω ε, πιστεύουμε ότι, επειδή και το λένε και τα δικαστήρια άλλωστε, όλοι οι μετανάστες έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δύσκολο ε, να θεσπιστεί ένα πλαίσιο τελικά που θα προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μεταναστών νομίμων και μη. Επίσης έχουμε τη σύμβαση του Διεθνούς ε, Γραφείου Εργασίας για τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας των οικιακών βοηθών. Ε, είτε είναι νόμιμη είτε όχι αυτή. Κάποιες χώρες ε, από το Βορρά βλέπουν ευνοϊκά με θετικό μάτι τη σχετική σύμβαση και επικυρώνουν. Άρα δεν είμαστε σαν διέξοδο. Τώρα, κέντρα φιλοξενίας. Και αυτό είναι ένα εργαλείο Τώρα το θέμα είναι γιατί χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται για ενημέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση, υγειονομική περίθαλψη κτλ. Τότε μπορεί να κάνει μεγάλο καλό. Εάν είναι ένα κέντρο κράτηση όμω, για να του ε, ε, κρατήσει εκεί αυτούς που μπαίνουν στη χώρα και μετά να τους ε, διώξει από τη χώρα αυτό δεν είναι θετικό. Για χερσαία σύνορο, Ουκρανία ε, δεν μπορώ να τα καλύψω όλα. Επικεντρώθηκα ε, στα σύνορα τα ελληνοτουρκικά και στη, στα σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Νησίας γιατί δεν μπορώ να καλύψω τα πάντα όπως είπα και βλέπω ότι είστε έτοιμος να με διακόψετε. Ολοκληρώνοντας λοιπόν θέλω να πω ότι το δικό μου έργο ουσιαστικά έγγειται στο να αλλάξω την, ε, το θεωρητικό πλαίσιο, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται Ακούμε πάρα πολλά πράγματα για, την, για τους μετανάστευση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αναδιατυπώσουμε τη γλώσσα αυτή και να τη βάλουμε σε μια προοπτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν μπορώ κι εγώ να συνεισφέρω σε αυτό, γιατί φυσικά μόνος μου δεν μπορώ να τα καταφέρω, αν συνεισφέρω θα έχω κάνει τη δουλειά μου. Ένα παράδειγμα. Διάκριση μεταξύ ε, smuggling, trafficking, ε, λαθρεμπόριο, διακίνηση. Πολλές φορές ε, ταυτίζονται αυτά τα δύο σαν να είναι το ίδιο κακά και τα δύο. Σίγουρα το λαθρεμπόρο, το smuggling είναι κακό, έχει σώσει και ζωές όμως. Αναρρυθμητοί μετανάστες έχουν χρησιμοποιήσει τους λαθρεμπόρους ε, για να βγουν από ένα δικτατορικό καθεστώς. Αυτό έγινε ε, κατά κόρον τον 20ο αιώνα. Μην μπερδεύουμε τα δύο πράγματα. Ε, δεν είναι το ίδιο η διακίνηση ε, και το ε, λαθρεμπόριο. Λαθρεμπόριο τσιγάρων, εντάξει, καλό είναι, αλλά δεν είναι τόσο όσο η διακίνηση, γιατί η διακίνηση είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το λαθρεμπόριο μπορεί να είναι κακό, αλλά μπορεί να σώσει και ζωέ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει λίγο ε, το ενοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο. Αυτό θα προσπαθήσουμε και εμεί να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Κρυπό, σα ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Άριας Φερνάντεθ,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 Ε, αναφέρθηκαν δύο μέλη τη Επιτροπή σα ε, στο Συμβουλευτικό Φόρουμ. Να σα πω πρώτον ότι ο ίδιο ο κανονισμό απαιτεί τη συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και για τη συγκρότηση του Συμβουλευτικού Φόρουμ και για, για τον ορισμό ε, των μελών ε, του Οργανισμού Θεμελιώδη Δικαιώματα. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Έχουμε λοιπόν ε, τη Συντακτική Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο. Έχουμε πρόσφατα ε, την εμπειρία ε, της συγκρότησης του Συνολευτικού Φόρουμ για τον ΕΑΣΟ. Χρειάστηκε 1,5 χρόνο για τη συγκρότηση αυτού του φόρουμ. Εμεί ελπίζουμε σε πέντε μήνε να έχουμε ολοκληρώσει αυτέ τι διαδικασίες. Η ετήσια συνεδρίασή μας γίνεται στο Σεπτέμβριο. Εκεί ελπίζω να τα καταφέρουμε, άρα δεν είναι τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον υπεύθυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα, θέλω να σα πω ότι εμεί δεν έχουμε μια τέτοια θέση, ούτε είχαμε όπως και πολλοί άλλοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ακολουθούμε τις ε, επιταγές πολιτικές, το, ε, είδαμε το 2011, θα ισχύσει και το 2012 και το 2013. Πρέπει να σεβόμαστε τον προπολογισμό, πρέπει να ζητήσουμε τροποποίηση του προπολογισμού μας για το 2012 από την αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή. Ελπίζουμε η τροπολογία αυτή να εγκριθεί μέχρι το Σεπτέμβριο, για να μπορέσουμε να ορίσουμε λοιπόν τον υπεύθυνο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλιώ δεν θα καταστεί δυνατό ούτε για φέτος. Σε ό,τι αφορά τι παραβιάσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ίσως θα ήταν ένα σκόπιμο να αναφέρω ότι οι υπάλληλοι αυτοί υπόκεινται στο εθνικό δίκαιο. Υπάγονται στις εθνικές αρχές, αυτοί τους ελέγχουν, σε αυτούς λογοδοτούν. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κοινέ επιχειρήσεις, στις 23 Μαΐου το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει, ε, θα ενημερωθεί και θα εγκριθούν τα σχετικά μέτρα σε περίπτωση ισχυρισμών για παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων απομακρύνεται ο σχετικός υπάλληλος και ενημερώνονται οι εθνικές αρχές και εφαρμόζονται τα ε, πειθαρχικά ή ποινικά μέτρα που προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Ακόμη και πριν ε, θεσπίσουμε τον κώδικα διοντολογία, στη νέα νομοθεσία και στον υπηρεσιακό κανονισμό υπήρχαν διατάξεις. Άρα, εάν υπάρξει κάποιο κρούσμα, μέχρι δεν είχαμε τέτοια περίπτωση, αν υπάρξει πάντως εφαρμόζονται οι σχετικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ο Γενικό Διευθυντή για την εντολή του, της Frontex, ε, το αφεντικό μα θέλετε, έκανε μία δήλωση. Έχουμε έλεγχο πάνω στους υπαλλήλους μας και γι' αυτό ε, θα εφαρμόσουμε πειθαρχικά μέτρα, εάν αυτό χρειαστεί. Και αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε ήδη πριν την έγκριση του κώδικα διοντολογίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Frontex για τον τρόπο με τον οποίο μας ε, αντιμετωπίζει η κοινή γνώμη, λυπούμε που το λέω, αλλά αν πραγματικά έτσι μας βλέπουν, εάν ε, έναν κέρβερο ε, στα σύνορα της Ευρώπης φρουρίου. Όχι, δεν είμαστε κάτι τέτοιο. οι συντονισμένες επιχειρήσεις της Frontex ε, σώζουν πολύ περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στον κόσμο. Άρα δεν είμαστε απλά ένας συνοριοφύλακας που κάνει έλεγχο στα σύνορα. Υπάρχει μια πολύ σημαντική ανθρωπιστική συνιστόσα. Έχουμε σώσει πολλού που κινδυνεύουν στη θάλασσα, για παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία μεταξύ Frontex και Εθνικών Κοινοβουλίων. Με τα λύπησα άκουσα ότι κλήθη Frontex να παραστεί και δεν συμμετείχαμε σε αυτή τη συνάντηση. Δεν το είχαμε ε, υπόψη. Λυπούμε. Έχουμε συνεχώς ε, επισκέψεις από εθνικούς βουλευτές και ε, μακάρι να έρθει και εκπρόσωπο του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Θα ελέγξω ε, την πληροφορία αυτή με το διευθυντή μου και θα δω γιατί δεν ήρθαμε ε, στην Πολωνία, γιατί δεν δεχθήκαμε τελικά την πρόσκλησή σας. Ε, νομίζω ότι έχω απαντήσει Νομίζω ότι έχω απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μη σας ανησυχεί αυτό που είπα, οι προσκλήσεις ε, που έμειναν αναπάντητες, σας τις αφήσουμε ως κάτι που πέρασε και στο ξεχάσουμε. Αλλά αυτό που έχω να πω τώρα είναι ότι αυτή η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να συμβάλλει στην οικοδόμηση της δημόσιας εικόνας της Frontex ως οργανισμού. Θα έλεγα ότι για αυτόν κυρίως το λόγο πρέπει να προωθηθεί μια τέτοια συνεργασία. Ο κύριος Τίμερμαν επίσης έχει αναφερθεί στο ίδιο ζήτημα. Η Frontex είναι ένας οργανισμός ε, διαχειριστικός. Και ε, δεν έχει δικές της ε, δυνάμεις καταστολής που προστατεύουν τα σύνορα. Τα σύνορα με επαφή με το Κοινοβούλιο μπορούμε να δούμε ποιοι είναι, μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιοι είναι οι σκοποί σας και το πεδίο εφαρμογή σας ειδικότερα μετά από την αλλαγή του κανονισμού της Frontex. Αυτό θα ήταν σημαντικό να δείξετε αυτή την όλη διαδικασία που είναι επικεντρωμένη στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι θα μπορούσατε να δείξετε ότι ο οργανισμός σας ε, σέβεται και αυτό το νέο πλαίσιο. Θα έλεγα ότι ο κύριος ε, Κρέπο ε, παρουσίασε δύο αξίες στη σημερινή συζήτηση την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών και τα δικαιώματα των μεταναστών αφετέρου, τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών. Πιστεύω ότι και οι δύο αυτές πτυχές ε, είναι θεμελιώδη σημασία. Το μόνο ερώτημα λοιπόν που πρέπει να απαντήσουμε είναι το πώς θα συμφιλιώσουμε αυτές τις δύο αξίες, πώς θα τις συμβιβάσουμε, την εθνική κυριαρχία και την προστασία των συνόρων με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για ένα ερώτημα μείζωνο σημασία και βέβαια ότι θα συνεχίσουμε να το συζητάμε στην, στην υποεπιτροπή μα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά του ε, προσκεκλημένους μας και θα ήθελα να ζητήσω τον να, την κυρία να ε, προεδρεύσει για τα επόμενα σημεία της ημερησίας διάταξη. Ευχαριστώ πολύ.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 Uh, Συνάδελφοι, να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει κάπως. Δεν φωνάζω αρκετά. Μήπως φωνάζετε εσείς πιο δυνατά από μένα. Σας παρακαλώ, όσοι δεν έχετε ε, αρμοδιότητα να είσαστε στην αίθουσα, τουλάχιστον να κάνετε ησυχία ή να βγείτε από την αίθουσα. Θα θυμάστε το θέμα... Έχουμε μάλλον μια ανταλλαγή απόψεων με τον Λουίς Γκουγέρεμο Περές Κάζας, που είναι Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τις εξελίξεις σε σχέση με την προηγούμενη ΝΤΑ το Τμήμα Μυστικών Υπηρεσιών της Κυβέρνησης της Κολομβίας. Θα θυμάστε ότι το θέμα αυτό είχε συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη το Μάρτιο και λόγω τεχνικών ε, προβλημάτων δεν ε, καταφέραμε να κρατήσουμε την τηλεφωνική επικοινωνία. Άρα λοιπόν ε, βάλαμε το θέμα αυτό στην σημερινή ημερήσια διάταξη και έχουμε την τύχη σήμερα να έχουμε τον κύριο Περές όχι μόνο σε τηλεφωνική επικοινωνία αλλά εδώ μαζί μας. Αυτό ασφαλώς θα μας δώσει καλύτερες δυνατότητες ε, για συζήτηση. Να προσκαλέσω και τον πρεσβευτή της Κολομβίας που και πάλι βρίσκεται μαζί μας σήμερα, όπως και την προηγούμενη φορά και όπως ε, ξέρετε, λόγω του θέματος, επειδή η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, συμμετείχε η ΝΤΑΣ θεωρεί ότι και το έργο μας στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα έπρεπε να παρακολουθείτε, γιατί δεν θέλουμε να υποστηρίζονται οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Γι' αυτό λοιπόν ο Πρόεδρος ζήτησε από την Αντιπρόεδρο Ιζαμπέλ Ντουράν να παρακολουθήσει το θέμα της ΝΤΑΣ και επειδή θα πρέπει σύντομα να φύγει από την ε, συνάντησή μας, δεν πρόκειται να προβώ σε κρεταμένες παρουσιάσεις. Θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην Ισαμπέλ για να μας ενημερώσει για το τι έχει πράξει ως τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Ιούλιο του 2011, αφού παρακολούθησα το φάκελο από το Βελίο μετέβη στην Κολομπή, βία για μια δεκαριά μέρες για να προσπαθήσω να αποκτήσω μια πλήρη εικόνα συνατώντα όλους τους ενδιαφερόμενους του φακέλου του ε, τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ενώσης, τον τύπο, τους πολιτικούς, ε, τους εκπρόσωπους της κυβέρνησης, τις διάφορες ενώσεις και ούτω καθεξής. Ε, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορείς να συναντήσει κανείς όλους και να προσπαθήσει να καταλάβει ποια ήταν η κατάσταση πριν από περίπου ένα χρόνο στην Κολομβία επί αυτού του φακέλου σήμερα 8-9 μήνες αργότερα έχω ακόμη πολλές ερωτήσεις για το θέμα. Σήμερα, παρότι εστάλησαν ωφέλιμα, πολύτιμα μηνύματα, όπως για παράδειγμα ένας νέος νόμος για τα θύματα, για την επιστροφή γεών, ένας νέος νόμος για τις μυστικές υπηρεσίες. Είχαμε μάλιστα εκείνη την εποχή την ευκαιρία να συναντήσουμε τον νέο διευθυντή της ΔΑΣ Τον παλιό, δηλαδή ο οποίο ασχολείται με τη μεταρρύθμιση του συστήματο. Ε, πιστεύω ότι παρόλα αυτά σήμερα, οκτώ μήνε αργότερα, εγώ έχω ακόμη πολλέ απορίε και κυρίω για μία από τι πτυχέ του φακέλου ε, την εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Βελγίου. Γιατί όπω γνωρίζετε, υπήρξαν υποκλοπέ, ε, email και τηλεφωνικών συνομιλιών και εδώ στο Βέλγιο στο πλαίσιο των στρατηγικών που χρησιμοποιούσε από αυτή την άποψη δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή που ζητήθηκε από τους Βέλγους δικηγόρους δεν καταφέρει ακόμη να μεταβεί επί τόπου ώστε να διεξάγει διερευνητική εξέταση για την επιλυσία αυτού του φακελού διότι πιστεύω ότι αυτός ο φάκελος θα πρέπει να επιληθεί ο ζήτημα αλλά πλήρως και επιλύοντας τα πάντα. Σήμερα λοιπόν εξακολουθώ να με καταλαβαίνω και πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να ασκήσουμε επιπλέον πίεση ώστε αυτή η Εξεταστική Επιτροπή να μεταβεί επί τόπου. Εξετάζοντας και τα άλλα ζητήματα όπως την ε, πρώην Διευθύντρια που εξορίστηκε στον Παναμά και διάφορους άλλους φακέλους θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε όσο γίνεται περισσότερο πριν αυτός ο φάκελο ντά ε, εξαφανιστεί στο πλαίσιο των αλλαγών που γίνονται αυτή τη στιγμή διότι με την παρέλευση των χρόνων ε, όταν αφήνουμε τα πράγματα ως έχουν τα αποδεικτικά στοιχεία θα εξαφανιστούν έτσι γίνεται σε όλες τις υποθέσεις πιστεύω λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να επιλύσουμε όλο αυτό το μυστήριο, όλο αυτό το ζήτημα είναι ένα μήνυμα που πρέπει να μας δώσει η Κολομβιανή κυβέρνηση. Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στο μέλλον, δεν ανακατεύουμε τις υποθέσεις της Κολομβίας από αυτή την άποψη, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να μας δώσει σημαντικά μηνύματα. Η Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να μεταβεί επιτόπου και να επιλύσει όσο το δυνατόν πιο πλήρως το φάκελο και το επαναλαμβάνω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσουμε σύντομα για μια συνθήκη ελεύθερη συναλλαγή με την Κολομβία. Υπάρχουν ε, διχογνωμίες, δεν είναι το ζήτημά μας βέβαια σήμερα αυτό, αλλά πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε μια τέτοια συνθήκη ανεξαρτήτως των εκατέρωθων θέσεων πιστεύω ότι θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμο να μπορέσουμε να λάβουμε από τις Κολομβιανές αρχές σαφή σαφείς ενδείξεις ε, για το γεγονός ότι ναι, μάλιστα συζητάμε αυτή τη στιγμή μια νέα συνθήκη, ωστόσο σα στέλνουμε κάποια θετικά μηνύματα όσον αφορά την επίλυση, την ολοκλήρωση από τα ανώτερα κλιμάκια αυτού του φακελοντά στο πλαίσιο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωση, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ουσιαστικά και τη Κολομβίας. Ολοκληρώνω λέγοντα ότι έχουν ε, γίνει κάποια βήματα αρχίζει ο φάκελος ε, να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη καθαρότητα τα διάφορα δηλαδή επίπεδά του διότι δεν μιλάμε για ένα απλό θέμα μιλάμε για μια ε, περίπλοκη υπόθεση που βάρει ε, σοβαρά κυρίως την σωματική ακαιρεότητα πολλών από τους συμμετέχοντες στην Κολομβιανή Δημοκρατία μια χώρα που υποφέρει από ζητήματα βίας είναι προφανέ αυτό. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε πολιτικέ εμπορικέ σχέσει με την Κολομβία με θετικό τρόπο, πιστεύω ότι εμεί ε, ω δημοκράτε ε, και ειδικά εμεί τα μέλη τη επιτροπή ΔΡΟΑ θα πρέπει να μπορούμε να δούμε καθαρά αυτό το ζήτημα, να υπεραμεινθούμε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. αυτό είναι ο στόχο μα η ανάγκη την οποία υπερασπιζόμαστε ω ε, βουλευτέ του Ευρωκοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση ώστε αυτή η Εξεταστική Επιτροπή με, εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Βελγίου, της Ισπανίας να μπορέσει να ρίξει φως σε αυτή την υπόθεση DAS πριν ξεκινήσουμε συζητήσεις το Σεπτέμβριο για αυτή την ε, συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κολομβίας. Αυτά είχα να πω σήμερα. Θα συνεχίσω να έχω αυτό το όραμα για τα πράγματα, διότι θεωρώ ότι η πολιτική αποτελείται από μηνύματα και αυτό το μήνυμα, ανεξαρτήτως των νομοθετικών μηνυμάτων που έχουν ξεκινήσει και των διαφόρων προβλημάτων της Κολομβίας, πρέπει οπωσδήποτε να επιληθεί από τους Κολομβιανούς. Εμείς ως Ευρωπαίοι έχουμε ηθικό καθήκον και σχετιζόμαστε άμεσα με αυτό το φάκελο, ε, ειδικότερα όσον αφορά τις υποκλοπές ε, των δικών μας μηνυμάτων και τηλεφωνικών συνομιλιών ε, εν αγνία μας. Θα πρέπει λοιπόν να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα ε, στέλνοντα αυτή την Εξεταστική Επιτροπή επιτόπου. Αυτά είχα να πω κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που θα χρειαστεί να σας εγκαταλείψω. Ωστόσο θα συνεχίσω να παρακολουθώ τις εργασίες της δικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνέχεια για αυτό το φάκελο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μείνουμε όλοι ενωμένοι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την επίλυση αυτού του φακέλου με σαφήνεια, καθαρότητα, δικαιοσύνη και ε, καταπολέμηση της ατιμορρησίας, ε, το βασικό πυλώνα της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ, Ιζαμπέλ. θα συνταξούμε και μια τελευταία έκθεση για αυτό το θέμα. Μπορείτε λοιπόν να το παρουσιάσετε και στη συνδιάσκεψη των Προέδρων. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο σε εσά, κύριε Πέρες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ε, υπενθυμίσω τη διάσταση των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί από μια υπηρεσία ασφάλειας και πληροφοριών του κράτους, η οποία παγόταν απευθείας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μιλάμε για πάνω από 600 θύματα. Μεταξύ αυτών υποστήρικτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, πολίτες, ε, αντιφρονούντες, ε, συνταγματικοί δικαστές, δικαστές στον ΟΤΑ του δικαστηρίου. Μιλάμε όχι μόνο για παράνομες ε, υποκλοπές, μιλάμε για δολοφονίες, μιλάμε για επανειλημμένες απειλές ε, κατά ε, θανάτου. Εδώ βλέπετε μία καμένη και διαμελισμένη και ε, χρωματισμένη με κόκκινο ε, στην κόρη ε, της Αντιπρόεδρου της Διεθνής Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι πρόεδρος του κολεκτίβου Δεαμπογάδος Χωσέ José Alvear Estrepo αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Οκτώ χρονών είναι η κορούλα της ε, κυρίας αυτής. Τη στείλαν αυτή την κούκλα για να δείξουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει η κόρη της αν συνεχίσει να προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στην αδελφό μου γιατί είναι γυναίκα και γιατί ε, κράτησε ε, ψηλά το λάβαρο αυτή τη μάχη παρά τι απειλέ που δέχθηκε. Σε ό,τι αφορά τώρα το, το δικαστήριο, νομίζω ότι είναι η μόνη χώρα η Κολομβία για την οποία οι πέντε δικαστές υπάρχουν, ε, για τους ε, δικαστές της οποίας αυτής οργάνωση υπάρχουν ε, προστατευτικά μέτρα, διότι τους απειλούσαν. Ποιοι τους έχουν απειλήσει αυτούς τους ανθρώπους. Όχι τρομοκράτες, παρότι έχουμε τέτοιες συγκρούσεις, αλλά από το ίδιο το κράτος δέχθηκαν απειλές οι δικαστές αυτές, από την υπηρεσία ασφαλείας, από την υπηρεσία μυστικών υπηρεσιών που παγόταν, όπως είπα, στον πρώτο της δημοκρατίας. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή ε, να θέσω τρία ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις και τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να απαντηθούν στο πέσο της συζήτηση. Πρώτον, έγιναν ό,τι ε, έγινε το απαιτούμενα ε, για να πάψουν οι κλιματικές ενέργειες ε, της Υπηρεσίας Μυστικών Υπηρεσιών της Κολομβίας. Δεύτερον, έχει τεθεί τέρμα στις παράνομες υπηρεσίες πληροφοριών. Τρίτον, Εμεί, υπέρ και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε εγγυήσεις και εχέγγυα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δέσμευσή μα, να προασπίζουμε τη ζωή. η ΝΤΑΣ πράγματι καθαρίστηκε την 31η Οκτωβρίου. Αυτό είναι γεγονός. Πάνω από 40 υπάλληλοι της ΝΤΑΣ έχουν πλέον ε, ε δικ, αντιμετωπίζουν ε, ε, είτε δίκες είτε πειθαρχική διαδικασία. Και ο κύριος Αλβάρο Ουρίμπεθ που ήταν πρόεδρος ε, πλέον καταδίκασε τον διευθυντή επειδή η υπηρεσία του ε, ουσιαστικά ε, ήταν υπεύθυνη για δολοφονίες και συγκεκριμένα για δολοφονία του καθηγητού Αλφρέδο Κορέα Δε Αντρέης. Καταδικάστηκε λοιπόν ε, ο Χορχέ Αουρέλιο Νογκέρα σε 25 χρόνια φυλάκιση. Υπάρχει όμως έλλειμμα δικαιοσύνης ε, απέναντι σε αυτά τα εγκλήματα. Πολύ σημαντικό έλλειμμα. Πολλοί υπάλληλοι της ΔΑΣ δέχθηκαν τι ε, ποινικέ τους ευθύνες ε, με κάποια συνεννόηση εκ των προτέρων. Αλλά έχουν πει στη Γενική Εισαγγελία ότι δεν θέλουν να μιλήσουν γιατί φοβούνται. Φοβούνται για τη ζωή τους και για τη ζωή των οικογενειών τους. και μάλιστα ένας κύριος ο οποίος κατέφυγε ε, στη ΣΥΠΑ ε, και το Δεκέμβριο μίλησε στη Γενική Εισαγγελία και είπε ότι φοβάται. Έχει γίνει ήδη αυτό δηλαδή. Τώρα, αν έχει τεθεί τέρμα στι παράνομε δραστηριότητε του Μέτρου Μυστικών Υπηρεσιών τη Κολομβία, δυστυχώ η απάντηση είναι αρνητική. Οι υπερασπιστέ ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όχι μόνο αυτοί, αλλά και πολλοί Κοινωνικοί ηγέτες εξακολουθούν να είναι θύματα διώξεων, διωγμών. Κάποιοι έχουν δολοφονηθεί ή έχουν απειληθεί. Ε, έχει απειληθεί η ζωή τους. Και πολλοί φεύγουν από τις περιφέρειες που ζούσαν και φεύγουν και από τη χώρα τους για να προστατευθούν. Ο ίδιος ο πρόεδρος Σάντος είχε καταγγείλει ότι υπήρχε ένα μαύρο χέρι πίσω από τα εγκλήματα των ε, ηθινόντων. Προσπαθούσαν να ανακτήσουν τις ε, γέες τους. Αυτό που δεν δέχθηκε ο πρόεδρος Σάντος παρόλα αυτά και όσο το δέχ, δεν το δέχεται νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να τον βοηθήσει σε αυτό το καθήκον ώστε να ξεφορτωθεί το μαύρο αυτό χέρι το κράτος, γιατί εξακολουθεί να βρίσκεται στα κρατικά γρανάζια αυτό το μαύρο χέρι και τον πιέζει τον ε, πρόεδρο. Και εμείς το καταγγέλουμε αυτό, το καταγγέλουμε στεναρά. Προσπαθεί η κυβέρνηση να μεταρρυθμίσει ε, το, το κράτος, κάτι που δεν τόλμησε να κάνει ο προηγούμενος πρόεδρος, ε, ο Άλβαρο Ουρίμπε. 30 χρόνια ε, έχουμε αυτό το καθεστώς που έχει στοιχήσει πολλές ζωές και προσπαθεί το, ο σημερινός πρόεδρος να αποκαταστήσει την συνταγματική τάξη Ξέρουμε ότι πολλοί ε, στρατιωτικοί έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δίκες που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε τις απαραίτητες διασφαλίσεις παρότι ο πρόεδρος ε, ε Σάντος ε, έκανε μία δήλωση για αφοπλισμό κάποιας οργάνωσης παρά το ότι πολλές φορές ε, ε μας επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια, νομίζω ότι είμαστε δυστυχώς, ε, ε, και είναι παράδοξο αυτό, σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι υπό τις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις του Αλβάρο Ουρίμπε. Ε, δεχόμαστε περισσότερες απειλές, ε, απειλές δέχονται υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολύ περισσότερες. Το 2011, 49 υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δολοφονήθηκαν στην Κολομβία. 26 ηγέτες ε, κοινωνιών, εκτοπιστέντων που έχουν ζητήσει τις ηγέες ε, τους δολοφονήθηκαν μεταξύ του 2010 και του 2011. Εμείς ε, εξακολουθούμε να μην εκφοβιζόμαστε παρότι παραβιάζονται, παρότι έχουμε βία κρούσματα, μας απειλούν ότι θα μας σκοτώσουν. Παρ' όλα αυτά οι έρευνες δεν προχωρούν, δεν βλέπουμε να ε, βρίσκονται ή να εντοπίζονται οι δράστες παρά τη δική μας ε, αποφασιστικότητα. Ολοκληρώνοντας, ε, θέλω να σας πω ότι θέλω να σας δείξω αυτή τη διαφάνεια για την επιχείρηση Ευρώπα. Επιχείρηση Ευρώπη, έτσι είχε ονομαστεί από την τότε ΝΤΑΣ. Επειδή είπατε ότι ανησυχείτε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομπία, σας δείχνω αυτό. Υπήρχε μια στρατηγική η οποία αναπτύχθηκε και είχε ως στόχο την εξουδετέρωση ουσιαστικά ε, του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Παράνομη δραστηριότητα η οποία επεκτάθηκε σε δεκάδες οργανώσεις ανάπτυξης και συνεργασίας, είτε ευρωπαϊκές, ε, αλλά όχι μόνο, και σε Ευρωπαίους πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κολομβία. Υπάρχει λοιπόν μια ποινική έρευνα που έχει ξεκινήσει στη χώρα αυτή, στο Βέλγιο, αλλά και στην Ισπανία και ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσει αντίστοιχη ποινική διαδικασία στη ΣΥΠΑ γιατί ε, διώχθηκαν πολίτες ε, Αμερικανοί μεταξύ άλλων. Ολοκληρώνω λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, με κάποιες ε, συστάσεις για να βοηθήσετε τον πρόεδρο Σάντος να ξεκαθαρίσει το κράτος για τη δημόσια δίκηση, να βγάλει αυτό το μαύρο χέρι, να το εξαφανίσει πριν την επικύρωση της ε, Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κολομβίας θα πρέπει να απαιτήσετε από το κράτος και από την κυβέρνηση της Κολομβίας ε, να καθαρίσει ε, τα αρχεία των στρατιωτικών πληροφοριών και τα αστυνομικά αρχεία. Να σβήσουν τα αρχεία, να καταργηθούν όλα αυτά τα αρχεία που έχουν φακελώσει του υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρέσβη γνωρίζει πολύ καλά τον δόκτωρα Ριμπέρα που ήταν υπουργό Άμυνα. Είναι στην ιστοσελίδα των ενόπλων δυνάμεων ακόμη. Λέει ότι εμείς κάνουμε νομικό πόλεμο ή πολιτικό πόλεμο, γιατί μας έχουν ε, μετατρέψει σαν στρατιωτικό στόχο. Αυτό πρέπει να πάμψει είναι θεμητός και ε, απαραίτητος για τη δημοκρατία ε, ο στόχος μας και το έργο μας. Εμείς επιμένουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει ένα τέλος πρέπει να σταματήσει ε, και να ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, για την κοινωνία. Πρέπει να σταματήσει η συνταγματική μεταρρύθμιση. Πρέπει να λάβει ένα τέλος η συνταγματική μεταρρύθμιση. Και θέλω τέλος να σας δώσω ένα μήνυμα. Το είπαμε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το είπαμε και στην Καγκελάριο και εγώ το επαναλαμβάνω εδώ. Εάν για την πρόσφαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν για τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει να καταπολεμήσουμε το έγκλημα, να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της ατιμορρησίας, για να έχουμε ένα κράτος δικαίου, για να έχουμε δημοκρατία, ε, για να έχουμε ε, πολιτική επίλυση της ένοπλης σύραξης ε, στην Κολομβία, για την ειρήνη. Εάν για όλα αυτά, αντί να, αυτά να αναγνωρίζονται, είτε μας σκοφαντούν, είτε μας δυσφημούν, είτε μας βάζουν στη φυλακή, εμείς παρόλα αυτά είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Η διεθνής κοινότητα, ο λαός της Κολομβίας, θα καταλάβει, πιστεύω, καλή αργά παρά ποτέ, θα καταλάβει ότι εμείς είμαστε αξιοπρεπείς, δρούμε με ευθύνη, υπευθυνότητα και ιστορική μάλιστα υπευθυνότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παρέσκά και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην EIS να μας πείτε τι κάνετε σε σχέση με την Κολομβία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να δώσουμε το λόγο πρώτα στον ε, πρεσβευτή της Κολομβίας σε πρώτη φάση. Ναι, ε, λυπάμαι, αλλά έχουμε κανόνες εδώ. Καταρχάς θα συζητήσουμε στο εσωτερικό της Επιτροπής και αν επιθυμεί στη συνέχεια ο πρεσβευτής θα πάρει το λόγο. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Σας ζητώ να πάρετε το λόγο. Ακολουθήσαμε το σκάνδαλο της ΝΤΑΣ από την αρχή. Ήταν πολύ σοβαρή η υπόθεση αυτή προφανώς. Μια υπόθεση την οποία θέσαμε κατευθείαν στη συζήτηση και στο διάλογο με την κυβέρνηση της Κολομβίας. Ένα θέμα το οποίο ανέκυψε σε διάφορες περιστάσεις σε ό,τι αφορά το διάλογο με τα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την κυβέρνηση. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που αναφέρθηκαν για τη σημασία του ρόλου των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της Κολομβίας, που, όπου τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Και γι' αυτό λοιπόν καλώς ορίσαμε τις δηλώσεις ε, που έγιναν από την ανάληψη των καθηκόντων του Πρόεδρου Σάντο σε ό,τι αφορά την προστασία των πρόσπιστων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι ήταν ξέσπασε το σκάνδαλο αυτό, ο Πρόεδρος Σάντος ε, ήταν υπουργό Άμυνα. Εκείνος λοιπόν ζήτησε να κλείσει η υπηρεσία DAS που είχε κατηγορηθεί για αυτές τις δράσεις. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του αυτό συνέβη και επίσης σημειώνουμε ότι διάφορες ε, έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από τους γενικούς εισαγγελείς και από τις δικαστικές αρχές όπου ασφαλώς στην Κολομβία όπου, όπως και αλλού ε, είναι ανεξάρτητες αρχές και φυσικά Χρειάζονται χρόνο οι έρευνες αυτές και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ασφαλώς να επιληθεί το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο αυτό, όπως αναφέρθηκε, αφορά εκατομμύρια υποθέσεις και σελίδες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να διερευνηθεί σε σύντομο διάστημα. Είναι σημαντικό λοιπόν οι φάκελοι αυτοί να κατασχεθούν από την εισαγγελία και από όσο γνωρίζω ε, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες ε, και κατά υψηλών αξιωματούχων που έχουν οδηγήσει σε καταδίκες όπως αναφέρατε. Καλωσορίζουμε ασφαλώς τις έρευνες αυτές και τις παρακολουθούμε και σχετίζονται άμεσα με τις κατηγορίες για δραστηριότητες εδώ, στην Ευρώπη και σε ό,τι αφορά την ίδια την υποεπιτροπή, να είστε βέβαιοι ότι το θέμα αυτό θα παραμείνει στην ημερήσια διάταξη των επόμενων μηνών. Μία υποσημείωση τώρα για το θέμα της δικαστικής μεταρρύθμισης και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα της παράτασης, την αλλαγή του καθεστώτος του συστήματος ε, στρατιωτικής δικαιοσύνης, το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με το ζήτημα που συζητάμε σήμερα. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο μας ανησυχεί και μας κάπως από την αρχή του ξεσπάσματος του σκανδάλου ζητήθηκε να μεταφερθούν τα θέματα αυτά, οι υποθέσεις αυτές στο κανονικό δικαστικό σύστημα, το οποίο και συνέβη εν μέρη. Τώρα εκφράζουμε ανησυχία για ενδεχόμενη παράταση της δικαιοδοσίας του στρατιωτικού δικαστηρίου ή ενδεχόμενη διεύρυνση της δικαιοδοσίας τους. Η κυβέρνηση έχει ζητηθεί αυτές τις μεταρρυθμίσεις επίσης να παραμεριστούν και στον διάλογό μας η κυβέρνησή μας, μας ε, η κυβέρνηση της Κολομβίας μας έχει αναφέρει ότι αυτό αποτέλεσε ε, αποτέλεσμα και της ευρωπαϊκής πίεσης. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και τώρα να ακούσουμε σχόλια, ερωτήσεις και παρατηρήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Κλούτε. Σας ευχαριστώ. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής, αλλά από την Επιτροπή μας, από την ομάδα μας, συγγνώμη, δεν υπάρχει άλλος αντιπρόσωπος δυστυχώς σήμερα, γι' αυτό λοιπόν ζητώ το λόγο και ασχολούμαι ασφαλώς με το θέμα της ε, Κολομβίας. Καταρχάς λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Περεσκάστα για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Νομίζω ότι στην παρούσα κατάσταση είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συζητάμε τα θέματα ε, Συμφωνίας ελεύθερου Εμπορίου που περιλαμβάνουν ε, ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άρα είναι σημαντικό να είμαστε ενήμεροι για την σημερινή κατάσταση. Η θέση της ομάδας μου είναι η εξής. Δεν θα πρέπει να υπογραφεί η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου όσο τα θέματα αυτά παραμένουν αναπάντητα και ιδιαίτερα αυτή η ιστορία με την DAS. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, κύριε Περεσκασάς, τοποθετηθήκατε ήδη, αλλά θα μπορούσατε να κάνετε κάποιες παραπάνω παρατηρήσεις για τη θέση αυτή του να μην υπογραφεί δηλαδή η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου προτού λυθεί το θέμα. Θεωρούμε ως ελάχιστη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να υπάρχει χωρίς όρους συνεργασία μεταξύ των Κολομβιανών και των Ευρωπαϊκών Αρχών και να συναυτούν συμφωνίες ε, δικαστικής και αρρωγής. Αυτή είναι η θέση μας. Οι βελγικές ε, αρμόδιες αρχές ε, ασχολούνται με τις κατηγορίες αυτές ε, υποκλοπής ε, και παρακολούθησης Ευρωπαίων βουλευτών και θα συμμετάσχουμε ασφαλώς στις ε, έρευνες αυτές. Αυτό ο σχόλιο από πλευρά της ομάδας μου. Θα ήμουν ευγνώμων λοιπόν αν θα μπορούσατε να μας κάνετε κάποιες διευκρινήσεις και κάποιες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Κλούτε. Ζητά κανείς άλλο το λόγο από τα μέλη της Επιτροπής. Αν όχι, Πρωτού δώσω το λόγο όμως ε, στον κύριο Πέρες για να απαντήσετε. Να πω ότι η κυρία Ριβέρα, εκπρόσωπος ε, της ε, Κολομπιανής Πρεσβείας, έχει ζητήσει το λόγο για τρία λεπτά. Όπως ξέρετε, έχει τρία λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μας δώσετε να μιλήσουμε για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τη δήλωση την πρόσφατη τη υπάτη εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για εξωτερικά θέματα και την πολιτική ασφάλεια. Τη δήλωση τη κυρία Άστον τη Δευτέρα Μαου τρέχοντο που ζητά την ε, άμεση και ανεφόρον απελευθέρωση του Γάλλου δημοσιογράφου Ρωμαίο Λαγκλουά, τον οποίον ε, πήγαγαν οι ΦΑΡΚ ε, πριν από δέκα ημέρες. Όταν παρακολουθούσε και κάλυπτε μια επιχείρηση των αρχών κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Για μια ακόμη φορά οι ΦΑΡΚ καταπιάζουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ανθρωπιστικό δίκαιο, για την πρόσπιση του αιματηρού παράνομου εμπορίου ναρκωτικών. Ο πρόεδρος Σάντος στη Σιγκαπούρη ε, είπε ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι και δεν μπορεί να είναι και ποτέ δεν θα είναι ε, κρατούμενη πολέμου. Επίσης θα ήθελα στη γραμματεία της Επιτροπής σας ε, να δώσω ένα έγγραφο το οποίο χθε έδωσα και στην πρόεδρο την κυρία Λόχ Μπίλερ με τις απαντήσεις της δηλώσεις της εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων το Μάρτιο. Ελπίζω έτσι να μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα την πραγματικότητα της Κολομβίας. Γίνονται κάποιες αναφορές σε ορισμένα από τα θέματα τα οποία είχε αναφέρει και ο κύριος Πέρης. Για το συγκεκριμένο ζήτημα της ΝΤΑΣ, τέσσερα σημεία. Πρώτον, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση, ο πρόεδρος Σάντος κράτησε την υπόσχεσή του να κλείσει την ΤΑΣ τον προηγούμενο Οκτώβριο η Γενική Εισαγγελία του κράτους, η Εθνική Αστυνομία και η Διοικητική Ειδική Μονάδα για την Μετανάστευση, πρόσφατα συσταθήσα μονάδα, ανέλαβαν τις σχετικές αρμοδιότητες. Φυλάσσονται όλα τα αρχεία της Γενικής, ε, του Γενικού Δικαιστικού Δικαστήριου της ε, Προκουραδορία Γενεράλ, που είναι ανεξάρτητο κρατικό όργανο. Επίσης υπάρχει ένας νέος νόμος πληροφοριών που ενισχύει την, ε, πληροφορία, τις πληροφορίες του κράτους. Υπάρχουν σαφείς περιορισμοί, απαγορεύσεις, διαφάνεια, σεβασμός των θεμελών και ελευθεριών. Υπάρχει μεταξύ άλλων κοινοβουλευτικός και δικαστικός έργο που προβλέπεται. Τρίτον, η κυβέρνηση στηρίζει και πολιτικά και δημοσιονομικά τη δικαιοσύνη και το διοικητικό δικαστήριο, την προκουραδορία για να ανακαλύψουν, να διαφωτίσουν την κατάσταση, για να τιμωρήσουν ε, υποδειγματικά, παραδειγματικά όλους τους υπεύθυνους για οποιαδήποτε παράνομη δράση. Μέχρι το Μάρτιο είχαμε λοιπόν 66 δίκες, 18 άτομα ε, μπήκαν στη φυλακή και 3 καταδικάστηκαν, μεταξύ αυτών και ένας πρώην διευθυντής ε, της υπηρεσίας. Τέλος, κάτι για τη δικαστική ανεξαρτησία. Η Κολομβία είναι κράτος δικαίου. Υπάρχει διάκριση εξουσιών και η Γενική Εισαγγελία και ο, ημέδιος, και για την ποινική έρευνα και οι δικαστές που κάνουν τις δικαστικές αποφάσεις είναι ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση. Είναι, υπάγονται στον νόμο και στις εγγυήσεις του ποινικού δικαίου, τις οποίες και σέβονται η κυβέρνηση σέβεται τη δικαστική ανεξαρτησία και αυτονομία που είναι σημαντικό στοιχείο της συνταγματικότητας, της αξιοπιστίας, της νομιμότητας στη χώρα μας. Περιμένουμε από τη δικαιοσύνη να δώσει τις απαντήσεις που μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να δώσει για όλα τα θέματα που έχουν καταγγελθεί. Τέλος και κατακλείδη η Κολομβία και η κοινωνία αλλά και οι διάφορες κρατικές οργανώσεις και φορείς έχουν αναλάβει αποφασιστική δράση ώστε να λάμψει ε, η αλήθεια δικαστικά για να αποδοθούν ευθύνες και για να υπάρξουν οι απαραίτητες συνταγματικές κανονιστικές αλλαγές για να μπορέσει να ε, πάψει η... το παρελθόν αυτό, το μαύρο παρελθόν να μην επαναληφθεί ποτέ. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Δίνω λόγο σε εσά, κύριε Περισκάσας, για να απαντήσετε την ερώτηση του κύριου Κλώτη. Και παρακαλώ να μην μιλήσετε περισσότερο από πέντε λεπτά, γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει τα χρονικά όρια. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, που είναι στη φάση της επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να πω συγκεκριμένα γι' αυτό ότι μια δημοκρατική ρήτρα έχει ενσωματωθεί στο κείμενο αυτής της ε, συνθήκης. Υπάρχουν δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και περιβαλλοντικά ζητήματα. Για μας πάντως εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία το ότι θα μπορούσε να επικυρωθεί μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών όσο στην Κολομβία συνεχίζουν να δολοφονούνται συνδικαλιστές, να δολοφονούνται αυτόχθονες ηγέτες, ηγέτες ε, των εκτοπιστέντων ή υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχει κανένα νόημα να επικυρωθεί μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και μετά να πει κανεί ότι ξέρετε, υπογράψαμε σύμβαση, ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με μια κυβέρνηση που εξακολουθεί να επιτρέπει σοβαρέ, βαρύτατε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο δυνατόν για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω το καλύτερο θα ήταν να βοηθήσετε τον πρόεδρο Σάντο να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται πριν την επικύρωση αυτής της ε, συνθήκης να τεθούν επιτάπητο κάποια θέματα, όπως αυτά που αναφέρα, ανέφερα και εγώ στην παρέμβασή μου. Θα πρέπει να γνωριστεί η νομιμότητα ε, του έργου των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει συκοφαντική εκστρατεία. Ε, δεν σταμάτησε αυτό μετά τον πρόεδρο Ουριμπέ. Συνεχίστηκε με τον πρόεδρο Σάντο η ίδια αυτή προσπάθεια συκοφαντικής δυσφήμισης πρώην Υπουργό Άμυνα και πρέσβη γνωρίζει πολύ καλά γιατί συζητούμε εμείς ζητήσαμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δημοσία να ανακαλέσει τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και της ε, Καγκελαρίου της Κολομβίας που το έργο της δικής μας οργάνωσης ε, Κολεκτήπο Τεποκάτος Χωσέ Αλβεάρ ρεστρέ σε μια δίκη που το δικηγόροι για πάνω από 16 ε, δικηγόροι προσπάθησαν να ε, καταδικάσουν και έγινε αυτό ε, 15 ετή δράση ε, του κράτους. Υπάρχουν αγνοούμενοι, υπάρχουν προσπάθειες να μας παρουσιάσουν εμάς ως διεφθαρμένους ότι εμείς χρηματιζόμαστε και πλουτίζουμε, ενώ ουσιαστικά θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας για να προασπίσουμε τις ζωές άλλων. Αυτό που μας είπε ο Πρόεδρος είναι ότι εγώ ποτέ δεν ανέφερα τη δική σας οργάνωση. Ποτέ δεν μίλησα για το κολεκτίβο Δεαμπογάδος, άρα δεν έχω να ανακαλέσω κάτι. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη το ίδιο είπε. Εγώ δεν μίλησα ποτέ για εσά, δεν σα ανέφερα ποτέ δεν ανέφερα κανέναν, κανένα μέλος της οργάνωσής σας, όμως η δημόσια κοινή γνώμη ε, ουσιαστικά στην ε, μάλλον δημόσια κοινή γνώμη παραμένουμε στιγματισμένοι. Η δραστηριότητά μας είναι μη κερδοσκοπική και πάντοτε εργαζόμαστε ακριβώ για να πάψει να υπάρχει αυτή η εξαθλίωση, να, πάψουν να υπάρχουν οι καταπιέσεις. Θέλουμε να συνεισφέρουμε σε μια μεγαλύτερη ε, διαφάνεια, συνταγματικότητα και καλύτερη υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε και να υπερασπιζόμαστε την ειρήνη. Ο κύριος Πρέσβης μίλησε για κάποιες έρευνες, ε, για κάποιους που μπήκαν φυλακή, για κάποιους που καταδικάστηκαν κτλ. Εγώ, κύριε Πρέσβη, σας ερωτώ να δεσμευτείτε να μας απαντήσετε εγγράφως, γιατί εμείς σας έχουμε επαναλημμένο θέσει το ερώτημα και στον ίδιο τον Πρόεδρο και στον Υπουργό Δικαιοσύνη και στον Υπουργό Άμυνας, γιατί μέχρι σήμερα ο κύριος Χωσέ Μιγγέλ Νταρμπάης, που ήταν υποδιευθυντής της ΔΑΣ και τον είχε ορίσει ο ίδιος ο πρόεδρος Άλβαρο Ουρίμπεθ, ο οποίος ε, δικάζεται για τρία πολύ σοβαρά εγκλήματα στην Κολομβία για τη δολοφονία ενός ε, ε, ε, γερουσιαστή, ενός δημοσιογράφου, για την απαγωγή μίας γερουσιαστού και δικάζεται και για όλα αυτά τα σχετικά με την τάσα. Γιατί μέχρι σήμερα ποτέ ο κύριος, μάλλον γιατί σήμερα εξακολουθεί να προστατεύεται από το στρατό και βρίσκεται ακόμη στην κατατίβαση στη στρατιωτική σχολή και προστατεύεται αυτός ο κύριος. Μήπως και καταλάβουμε τελικά. Ε, ε, μήπως εξακολουθεί να υπάρχει καθεστώς τρόμου στη χώρα μας. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Περέσκά σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Όπως είπαμε στην αρχή, θα αναφέρουμε μέσω της κυρίας Διουράων στη συνδιασκέψη των Προέδρων όπως κατάλαβα από τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η ΕΕΣ και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρισκόνται επί τόπου ε, παρακολουθούν στενά πολύ σοβαρές περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν θέλετε να υποβάλλετε γραπτές δηλώσεις, παρακαλείστε να το πράξετε. Ευχαριστούμε πολύ και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, και καθώς ε, ε, θέλουμε να διατηρήσουμε την ημερομία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, παρακαλώ όσοι αναχωρήσετε, τώρα που θα αλλάξουμε θέμα, να αναχωρήσετε σε... χωρίς φασαρία. Το επόμενο θέμα μας λοιπόν αφορά την κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Με ενημέρωσαν ότι πολλοί από εμάς ε, γνωρίζουν ότι πολλές είναι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία και παρόλα αυτά σπάνια τι συμπεριλαμβάνουμε στην ημερήσια διάταξή μας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να ξεκινήσω και θα αποφασίσουμε στο τέλος της συζήτησης τη συνέχεια αυτού του θέματος και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε. Η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη μεγάλη Ισλαμική χώρα που δεν έχει επικυρώσει τις δύο μεγάλες συνθήκες ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα πολιτικά δικαιώματα και για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Είναι μία από τις λίγες χώρες, από τις ελάχιστες μάλιστα χώρες που δεν ψήφισε υπέρ το 1948 ε, όταν υιοθετήθηκε η Παγκόσμια Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Έθνη το 2009 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά την παγκόσμια περιοδική αναθεώρηση, μια διαδικασία κατά την οποία οι διαφορές κυβερνήσεις συζητούν τι είδους βελτιώσεις ε, ή τι επιδεινώσεις έχουν ε, παρατηρηθεί. οι αρνητικές εξελίξεις έχουν λάβει χώρα. Υπήρξε ένας μεγάλος κατάλογος, όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε μπορείτε να το διαβάσετε σε αυτό το UPR του 2009 όπου η Σαουδική Αραβία παραδεχθήκε επίσημα ότι πρέπει να βελτιώσει σημαντικά και να υλοποιήσει τις συστάσεις άλλων όπως και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το απέτησαν για παράδειγμα ε, κατάργηση ή περιορισμό της θανατικής ποινής ε, και κατάργηση της ε, ανδρικής κυδαιμονίας των γυναικών. Θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Βίλκη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί αυτές οι συστάσεις. Ε, σας υπενθυμίζω επίσης ότι το Φεβρουάριο στο κοινοβουλίο μας ε, μάθαμε ότι η κυβέρνηση της Μαλαισίας ε, πέστειλε πίσω στη χώρα του έναν πολιτή της Σαουδικής Αραβίας λόγω κατηγοριών αποστασίας ουσιαστικά αλλαξοπιστίας Αλλαξοπίστηση στο οποίο στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες μουσουλμανικές χώρες ε, θα υποστεί θανατική ποινή. Υπήρξε λοιπόν διεθνής ε, διαμαρτυρία κατά αυτή της απόφασης της μαλαισιανής κυβέρνησης και ο πρόεδρος μας, ο κ. Σούλτς, ε, στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου είχε ζητήσει υπεύθυνα να μην σταλεί πίσω στη χώρα του Απέτυχαν όμω όλα αυτά και ο ελληνικό άνθρωπος βρίσκεται πίσω στη Σαουδική Αραβία. Υπογραμμίζω ξανά ότι απαιτούμε έντονα να μην εκτελεστεί. Επίσης υπέγραψα εγώ μια επιστολή για αυτή την υπόθεση. Συνυπέγραψα την επιστολή με μια διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Αραβική Χερσόνησο. Στείλαμε την επιστολή αυτή στον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας ε, στην Βρυξέλλες στις 15 Μαρτίου αναφέρω λοιπόν ένα κομμάτι σας διαβάζω τώρα ένα κομμάτι της απάντησής του η ελευθερία γνώμης στη Σαουδική Αραβία και στο βασίλειο αυτό διασφαλίζεται και είναι ευπρόσδεκτη στο πλαίσιο της, ε, του σεβασμού της θρησκείας η παρέτηση από ε, άλλες θρησκείες υπέρ του Μωάμεθ. Ε, η διακομόδηση του Μωάμεθ αποτελεί έγκλημα στο βασιλειό μας. Ε, όλοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν σεβασμό προς την Ισλαμική θρησκεία. Αυτό καθιστά σαφές ότι δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την περίπτωση του κ. Κασκάλη. Για να συζητήσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Σαουδική Αραβία, καλώ ορίζω εσά, κύριε Κρίστοφ Βίλκε, ερευνητή του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και επειδή έχουμε μεγάλο κατάλογο, συμφωνήσαμε να επικεντρωθείτε σε ορισμένες από τι σοβαρέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται υποκράτηση, που έχουν κατηγορηθεί και φυλακιστεί από το Δικαστήριο ασφαλέία της Σαουδική Αραβίας όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και των θρησκευτικών μειονοτήτων. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε και θα ακούσουμε και την άψη τη ΙΕΕΣ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε και κύριοι. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε ένα σημαντικό ιστορικό σταυροδρόμι. Ε, μεταβάσεις μεταξύ γενεών ε, έχουν ως αποτέλεσμα κρίση στην κυβέρνηση και στην πολιτική συμμετοχή. Η κυβέρνηση της Σαουδικής ε, Αραβίας αντιμετωπίζει αυτές τις κρίσεις ενώ οι αυξανόμενες απαιτήσει για το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζονται με έλλειψη ανοχής και καταστολή. Ο βασιλιάς που πέθανε πέρυσι ήταν νέος και ο νέος πρίγκιπας βρίσκεται, είναι άνω των 70 ετών. Η μετάβαση σε μια ηγεσία τρίτης γενιάς διαδόχων του βασιλιά Αμπτουλαζίζ ε, έχει ανασταλεί εδώ και κάποια χρόνια. Στο μεταξύ, 60% του πληθυσμού της χώρας των 90 εκατομμυρίων είναι κάτω των 18. Δεκαετίες πολιτικής ε, αντικατάστασης ε, των μεταναστών εργαζομένων ε, με κατοίκους Σαουδικής Αραβίας καθυστερούν διότι θέλουν υψηλότερους μισθούς και δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι. Η κατάσταση για τις γυναίκες είναι ακόμη χειρότερη. Ο βασιλιάς Αμπταλάχα έχει επενδύσει για τη δημιουργία βιομηχανικών και οικονομικών πόλεων σε όλο το βασίλειο και για επιστημονική εκπαίδευση ώστε να διαφοροποιήσει την οικονομία από το πετρέλαιο και να θέσει τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη. Ωστόσο, οι αλλαγέ για μια κοινωνία που θα σέβεται περισσότερα δικαιώματα θα προελθεί από την νέα γενιά, η οποία ελπίζω θα μπορέσει να επηρεάσει θετικά τη χώρα σε αυτό το σταυροδρόμι. Οι νέοι οδηγούν τι αλλαγέ ε, στη χώρα αυτή μέσω τη χρήση του διαδικτύου, όπου αποκτούν νέε μορφέ επαφή, έκφραση και επιχειρηματικότητα. Πριν από 7 χρόνια, όταν ξεκίνησα, συχνά συνομιλούσα με πολλούς μεταρρυθμιστέ, νέους ε, Άραβε, ε, οι οποίοι δημοσιεύουν σήμερα τι απόψει του στο Twitter. Όσον αφορά την πολιτική συμμετοχή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κυβέρνηση καθυστερεί, ενώ οι νέοι χαράσουν νέε ελευθερίε από μόνοι του. Ε, και η κυβέρνηση περιστασιακά τις αποδέχεται. Υπάρχουν τρία θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα αναφερθώ και στις θρησκευτικέ μειονότητες που πιστεύω είναι σημαντικές ε, για τη διασφάλιση των τριών ελευθεριών ε, ε, ελευθερίας άποψης δικαστηρίου και των γυναικών. Η Σαουδική Αραβία έχει μια πολύ ενεργό κοινότητα στο Twitter τελευταία στη Σαουδική Αραβία οι ηθοποιοί ε, διακομωδούν την κυβέρνηση σε ιδιωτικέ συνεδριάσει. Υπάρχουν αυτέ οι πτυχέ τη Σαουδική Αραβία που γνωστά δεν είναι γνωστέ. Όλα αυτά γίνονται παρά τι κυβερνητικέ πολιτικέ. Τα τελευταία πέντε χρόνια η Σαουδική Αραβία έχει ε, ψήφισε πιο αυστηρού νόμου για την ελευθερία έκφρασης ε, το 2007 ψήφισε ένα νόμο κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που χρησιμοποιήθηκε πριν από ένα μήνα για την καταγγελία ειρηνικών αντιφρονούντων. Τον Ιανουάριο του 2007 η Σαουδική Αραβία ρύθμισε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που απαιτούν, απαιτώντας άδειες για τις νέες ιστοσελίδες και ουσιαστικά καταργώντας τις δυνατότητες, ελέγχοντας όλες τις επικοινωνίες ε, και όλα τα μηνύματα. Τον Απριλίο του 2011 ε, επέκτηνε την εφαρμογή του τρέχοντος νόμου για τις δημοσιεύσεις και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και έτσι περιόρισε τις δημοσιεύσεις καθιστώντας το εγκληματικό το να δημοσιεύει οποιοδήποτε οτιδήποτε κατά του βασιλιά ή της θρησκείας. Ε, ακούσαμε ότι σχεδιάζεται ακόμη μεγαλύτερος περιορισμός όλων αυτών των δικαιωμάτων. Παρότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα το 2010, ο βασιλιάς Αμπτουλάχ περιόρισε τη λήψη αποφάσεων σε ε, ιερείς ε, στο πλαίσιο της κυβέρνησης. Συνεχίστηκαν συνεχίστηκε ε, το μπλοκάρισμα ιστοσελίδων εντός του Βασιλείου και ελάχιστες υποθέσεις παραβίασης του νόμου περί δημοσίευσης γίνονται δημόσιες. όλες, μας, ε, όλες οι προσπάθειες ελευθερίας άποψης αντιμετωπίστηκαν με ε, αυστηρότητα. Ζητήθηκαν πρόσφατα εκλεγμένο κοινοβούλιο. Υπήρξε μια ομάδα που θέλησε να δημιουργήσει το πρώτο πολιτικό κόμμα και στο facebook ε, έχουμε το site Date of Rage. Οι γυναίκες προσπάθησαν να οδηγήσουν. Η κυβέρνηση άφησε όλους αυτούς τους τους ετούντες μόνους τους. Όλοι ε, όσοι ανακρίθηκαν δήλωσαν ότι δεν θα ξαναπράξουν κάτι παρόμοιο εκτός από έναν ο οποίος καταδικαστήκε σε θάνατο. Το Day of Rage, οι Σαουδικές Αρχές και όλοι οι κληρικοί απαγόρευσαν οποιασδήποτε διαμαρτυρίες, είτε ειρηνικές είτε όχι. Ω αποτέλεσμα, κανένα δεν κατεβήκε στου δρόμου εκτό από έναν ο οποίο συλλήφθηκε διότι μίλησε στο BBC. Ένα άλλο άτομο που δημοσίευσε ένα βίντεο online ήταν ε, συλλήφθηκε και οι δύο παραμένουν κρατούμενοι και θα δικαστούν για την ειρηνική τους διαμαρτυρία στην Ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας όπου ζουν περίπου 2 εκατομμύρια ΣΥΙΤΕΣ. Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν το Φεβρουαρίο συνέξαν, χωρίς διακοπή. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν συλλάβει εκατοντάδες όπως και του ποιητή Αλεμχατίκ, ο οποίος παραμένει, καθώς και ηγέτες των ΣΥΙΤΟΝ που παραμένουν κρατούμενοι. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν σκοτώσει πάνω πολλούς ε, συζητές ε, υπό συνθήκες αδιευκρίνηστες. Μικρές διαμαρτυρίες από συγγενείς ε, κρατουμένων χωρίς δίκη έχουν λάβει χώρα το Μάρτιο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο αποτέλεσαν, εμπνεύστηκαν από ε, τις αραβικές εξεγέρσεις ε, στον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι οργανισμοί υπερασπίσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Υπάρχει μία ομάδα, Saudi Civil and Political Rights Association, που ξεκίνησε το 2009. Οι ιδρυτές της, ε, ειδικότερα ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ε, του έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία, απειλείται και έχει κληθεί στο γραφείο του εισαγγελέα πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες η Αντάλα. Μια νέα οργάνωση από το Φεβρουάριο του 2012 δεν έχει λάβει καμία απάντηση όσον αφορά το αίτημά τη για κυβερνητική άδεια. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει νόμους για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Στο δικαστικό σύστημα οι μεταρρυθμιστές, οι ΣΥΙΤΕΣ όλοι συμφωνούν για μια προτεραιότητα ε, τη δίκαιη δίκη για εκατοντάδες κρατούμενους που έχουν συλληφθεί ε, στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής ε, νομοθεσίας από το 2003. Το 2008 δημιουργήθηκε ένα δικαστήριο αντιτρομοκρατικό. Πολλοί κατηγορήθηκαν, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν σε, και κλεισμένων των θυρών και χωρίς δικηγόρους ή ορισμένες φορές ε, με πολύ συγκεκριμένους δικηγόρους και χωρίς ε, ελευθερία επιλογής. Ε, το 2011 ήδη δικάζονται οι ειρηνικοί αντιφρονούντες καθώς και επικριτές ε, του θρησκευτικού εξτρεμισμού. Το 2007 ο βασιλιάς Αμπτουλά ξεκίνησε μεταρρυθμίσεις δίνοντας μεγαλύτερη ανεξαρτησία στο δικαστικό σώμα, ε, έδωσε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση. Ο οργανισμός ΑΚΠΡΑ της Σαουδικής Αραβίας χρησιμοποίησε το διοικητικό δικαστήριο για να υποβάλει πολυάριθμες εφέσεις για αυθαίρετη κράτηση και βασανιστήρια. Συνεχίζει ωστόσο να μην υπάρχει καμία υπευθυνότητα για ε, λογοδοσία για τα βασανιστήρια. Έχουν υπάρξει τρεις γνωστές περιπτώσεις ε, για ομολογίες ε, όπου έχουν αποκομιστεί μέσω βασανιστήριων από φυλακισμένο όπως οποίος υπέστη ακροτηριασμό ποδιού. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ένα σημείο για το ποινικό δίκαιο. Ότι δεν υπάρχει ποινικό δίκαιο, δεν υπάρχει κώδικα ποινική δικονομία στη Σαουδική Αραβία που να αναφέρει ποιο ακριβώ είναι το έγκλημα. Οι εισαγγελεί και οι δικαστέ ε, καθορίζουν το έγκλημα ανάλογα με την πράξη. Και δεν υπάρχει νομικό ορισμό των εγκλημάτων. Οι Σαουδάραβες κατηγορούνται γιατί έχουν πολύ μακριά μαλλιά ή κλέβουν σε ένα ε, διαγώνισμα ή δεν υπακούν τους γονείς τους. Όλα είναι ανοιχτά προς τη διερμηνία. Η διακομόδηση του Ισλάμ δεν γράφεται πουθενά ως παραβίαση του νόμου στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για ερμηνεία. Αυτό επεκτείνεται και στα οικογενειακά ζητήματα. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ακουστεί υποθέσεις για υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναγκάζονται να διαζευθούν από τις γυναίκες τους διότι λένε ότι είναι άπιστοι χθες ένας ακτιβιστής υπέστη ε, απαγόρευση κυκλοφορίας των... ενώ ήθελε να συμμετέχει σε, μια, σε ένα συνέδριο στις Ηνωμένες αυτή τη στιγμή αναγκάστηκε να χωρίσει τη γυναίκα του και κρατείται. Τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν πολύ εμφυλεγόμενο ζήτημα. Άκουσα σε πολλές περιπτώσεις από φίλους ε, ε, του Βασιλείου ότι η Σαουδική Αραβία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η πιο ε, γνωστή ε, μεταρρυθμίση ήταν το 2011, το Σεπτέμβριο, για πολιτικά δικαιώματα, όπως δήλωσε ο Βασιλιάς. προκειμένου να έχουν δικαίωμα εκλέγην και εκλέγεστε στις κοινοτικές εκλογές. Ας κοιτάξουμε τις κοινοτικές εκλογές και τις δημοτικές εκλογές. Το Σεπτέμβριο του 2011 λοιπόν έγιναν εκλογές τέτοιες. Από τα 90 εκατομμύρια Σαουδάραβες, 60% είναι 118. Άρα έχουμε 5 εκατομμύρια Και ήταν πάρα πολύ λίγοι τελικά αυτοί, 35.000 αυτοί που πήγαν στις ε, κάλπες, που προσήλθαν στις κάλπες. Οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία προφανώς έχουν χαμηλότερη ποσοστό προσέλευσης. Άρα στις μελλοντικές εκλογές θα είναι πάρα πολύ μικρή η αριθμή των γυναικών κάτω των 75.000 που θα προσέλθουν στις κάλπες. Είναι καλή η συμβολική σημασία της ε, κίνησης, ε, αλλά μην περιμένουμε και σπουδαία πράγματα. Επίσης, ο Βασιλιάς ε, ανοίγει την αγορά εργασίας στις γυναίκες. Είναι 15% η εκπροσώπηση των γυναικών σήμερα. Αξιέπαινο λοιπόν, ε, αξιέπαινη η πρωτοβουλία του. 330.000 ε, και πλέον είναι οι γυναίκες στη ε, Σαουδική Αραβία που έχουν ψηλές υψηλού επίπεδου σπουδέ, αλλά δεν έχουν δουλειά. Τετραπλάσιο τα ποσοστά ανεργία στις γυναίκες και 60% ωστόσο των γυναικών, των φοιτητών στο πανεπιστήμιο είναι γυναίκες. Ζητείτε για παράδειγμα στα καταστήματα με για εσώρουχα να μην ε, δουλεύουν άνδρες αλλά γυναίκες. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2005 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τόσο πολύ καιρό παίρνει ακόμα και μια, ακόμα και μια τόσο μικρή πρωτοβουλία. Τα βασικά ζητήματα για τις γυναίκες έχουν μείνει απαράλλακτα ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την ανδρική κυδαιμονία. Παρά τις δεσμεύσεις που αναλήφθησαν, δεν έχει γίνει α, ιδιαίτερη πρόοδος. Ακόμα οι γυναίκες δεν μπορούν να βάλουν ξενοδοχείο μόνες τους. Χρειάζονται ε, άδεια από άντρα της οικογένειάς τους για να μπορέσουν να πάνε σε ένα ξενοδοχείο, να σπουδάσουν, να βγουν έξω σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, ίσως να είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής ε, έναντι των γυναικών. Η Human Rights Watch ε, δημοσίευσε σχετική έκθεση πρόσφατα, από την οποία ε, προκύπτει ότι ουσιαστικά δεν επιτρέπεται η συμμετοχή γυναικών σε αθλητικές δεν υπάρχουν ε, αθλητικές λέσχες στις οποίες να συμμετέχουν γυναίκες και το 2009-2010 και το Φεβρουάριο του 2012 ε, η κυβέρνηση έκλεισε ε, γυμναστήρια για γυναίκες. Και φυσικά στην Ολυμπιακή Αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας δεν προβλέπεται γυναικεία συμμετοχή και ακόμα και αν κάποια γυναίκα προσκληθεί προσωπικά θα πρέπει να έχει και δαιμόνα άντρα για τις παραβιάσεις ε, των θρησκευτικών δικαιωμάτων. Γίνονται ε, κατηγορίες, ακούμε κατηγορίες για την ε, διακριτική μεταχείριση των χριστιανών, των σιητών στην αγορά εργασία, στη δικαστικό σύστημα, σε ό,τι αφορά την ελεύθερη έκφραση και άσκηση της θρησκείας του. Θεωρώ λοιπόν, συνοψίζοντας, ότι υπάρχει κάποιος, ε, ε, κάποιο περιθώριο για την... Υπάρχουν ελπίδες για τη Σαουδική Αραβία, δεδομένης και της δημογραφικής κατάστασης στη Σαουδική Αραβία, αλλά ας μην είμαστε υπεραισιόδοξοι σε ό,τι αφορά όσους θέλουν γρήγορη εφαρμογή των ε, κανόνων για την προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Πιο γρήγορα κινείται η κοινωνία των πολιτών στη Σαουδική Αραβία παρά ε, ο νόμος. Λέει λοιπόν η Σαουδική Αραβία ότι δώστε μας χρόνο και θα κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, δεν το αμφισβητώ αυτό, αλλά θεωρώ ότι η ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων αυτών δεν ε, είναι στο ύψος των όσων περιμένει η κοινωνία. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, για την πολύ λεπτομερή αυτή παρουσίαση που καταδεικνύει ότι όντως υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Να καλέσω τον Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον κύριο Κοζίνη, να πάρει το λόγο. Είναι υπεύθυνο ε, για το Συμβούλιο για την συνεργασία με τον ε, Περσικό Κόλπο και τον κύριο Αντώνη Αλεξανδρίνη. Ίσως θα μπορούσατε να μοιραστείτε το χρόνο που έχετε. Ο κύριος Μπουσίνη καταρχάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βίλκε. Και για την παρουσίαση του αυτή. Όπως ως υπηρεσία εξωτερικής δράσης ασφαλώς συμφωνούμε με πολλές από αυτές τις ε, πλευρές. Ελπίζουμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα να τεθούν άμεσα τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας όσο το δυνατόν συχνότερα, γιατί όπως ξέρετε έχουμε μία αντιπροσωπεία στη Ριχάτ και βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο παρά το γεγονός ότι δεν δίνεται δημόσια διάσταση. Πάντα όμως βρισκόμαστε σε διάλογο για τα ζητήματα αυτά με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Τι μας ανησυχεί ιδιαίτερα, καταρχάς, η εφαρμογή τη θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο συχνά θίγουμε. Μα ανησυχεί ιδιαίτερα το υψηλό ποσοστό εκτελέσεων και καταδίκη στην Σαουδική Αραβία. Συμπεριλαμβανομένων και καταδικών για εγκλήματα τα οποία δεν θεωρούνται συνήθως ιδεχθεί. Ε, Είναι ανησυχητική αυτή η τάση, θεωρούμε, των θανατικών καταδικών. Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι η ελευθερία έκφρασης. Και τρίτον, θα ήθελα να τονίσω το θέμα της ελευθερίας ε, της ανεξιθρησκείας και της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων. Όλα αυτά τα ζητήματα διαρκώς συζητιόνται και με τις αρχές της αυτικής Αραβίας και με το σύνολο των χωρών του Περσικού κόλπου θα ήθελα να σας υπενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι πρόσφατα στα τέλη Μαρτίου έγινε η ετήσια συνάντηση των υψηλών αξιωματούχων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Περσικού κόλπου. Και ορίστηκε και ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκφράσαμε τις ανησυχίες μας ε, και εκφράσαμε και τα ζητήματα που μας απασχολούν. Πρέπει να πω ότι η συζήτηση ήταν πολύ ειλικρινής, ανεκτή και έντονη. Αυτό το θέμα τακτικά εμφανίζεται στις συναντήσεις που έχουμε στα ανώτερα επίπεδα, σε υπουργικό επίπεδο. Πέρσι το, στο Αμπουντάμπι τον Απρίλιο έλαβε χώρα η τελευταία τέτοια συνάντηση και στην ε, περίσταση αυτή τέθηκε ένα θέμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συζητήθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συνοψίζονται και σε μία κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στα τέλη της συνεδρίασης. Και ασφαλώς και θέλουμε τα θέματα αυτά να τα συζητήσουμε και με τις έξι χώρες του Περσικού κόλπου, αλλά και με το Συμβούλιο για τη Συνεργασία στον Περσικό κόλπο. Στην επόμενη Υπουργική Συνάντηση που θα λάβει η χώρα, ελπίζουμε σε λίγες εβδομάδες, επιπρόσθετα σε ό,τι αφορά την Σαουδική Αραβία. Θα ήθελα να τονίσω ότι με το γραφείο μας στο Ριχάντ προσπαθούμε να λάβουμε πληροφορίες για διάφορες μεμονωμένες υποθέσεις, όπως αναφέρθηκε. Αλλά πολλές είναι αυτές οι υποθέσεις που προσελκύουν την προσοχή μας. και το Κοινοβούλιο μέσω ερωτήσεων. Εμείς πάντα προσπαθούμε να συζητάμε τα θέματα αυτά με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας και να πω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις καταφέρνουμε να διεξάγουμε διάλογο. Δεν σας κρύβω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο διάλογος αυτός δεν είναι ο ευκολότερος δυνατός. Αλλά τουλάχιστον καταφέρνουμε να μοιραστούμε τις ανησυχίες μας με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Συνολικά πρέπει να σας πω ότι αυτό εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό τμήμα των σχέσεων μας με την Σαουδική Αραβία αλλά και με όλη την ομάδα των χωρών του κόλπου. Και ασφαλώς και θα συνεχίσουμε τη δράση αυτή στο μέλλον και θα λάβουμε όλα τα μέτρα τα οποία θα κρυθούν απαραίτητα ή δέοντα. Θα ήθελα... Δεν ξέρω αν θα θέλει ο συνάδελφος κάτι να προσθέσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Γουίλκε για την πολύ ακριβή παρουσίαση. Ο προλαλής σας συνάδελφος ε, σας και αγράφησε την πολιτική μας απέναντι στην ε, κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία. Θα ήθελα να πω ότι και στις δεμερείς επαφές που έχουμε αλλά και σε επαφές Ευρωπαϊκής Ένωσης GCC θέτουμε συνεχώς ε, πάγια τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, σε ατομική βάση και γενικά. Αναφέρατε τον κύριο Κασκάρη. τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο κύριος ε, Κασκάρη δεν αντιμετωπίζει θανατική ποινή πλέον, διότι φαίνεται ότι μετανόησε και κατά πάσα πιθανότητα θα υποβληθεί σε μία ελάσσονα ποινή. Με βάση τελευταίες ε, πληροφορίες είναι σε κατοίκον κράτηση οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας επιμένουν σε αυτό γιατί λένε ότι είναι για τη δική του προστασία. Ε, ε, ένας άλλος ε, αντιφρόνο, ένας άλλος μάλλον ο οποίος αντιμετωπίζει ε, κάποιες κατηγορίες για την ημέρα της αγανάκτησης και ο κύριος Αλμπατζάντη που αναφέρατε και για τους Ιήτες και την Ανατολική Επαρχία. Θέλω να σας πω ότι όλες αυτές ε, τις υποθέσεις και όλες αυτές τις ανομικές περιπτώσεις παρακολουθούμε και τους σύναγκες και είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τις αρχές ε, και ε, στην αντιπροσωπεία μας στο Ριάντ και παρακολουθούμε καθημερινά την κατάσταση. Ήθελα να προσθέσω ότι σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, εμείς ενθαρρύνουμε τις ε, αρχές της Σαουδικής Αραβίας να επικεντρωθούν στα παραδοτέα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, αναθεώρηση του UPR. Πριν από τρία χρόνια δέχτηκε η Σαουδική Αραβία μία δέσμη συστάσεων. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τη χώρα να εφαρμόσει τις συστάσεις αυτές που θα μπορούσαν να εστιάζουν κυρίως στην δυνάμωση των γυναικών, στην ελευθερία του συνεταιρίζεστε, του συνέρχεστε και την ελευθερία έκφρασης. Είπατε ότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει και πολύ blogging ε, μετά την Αίγυπτο είναι η δεύτερη χώρα με τα περισσότερα blogs η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τι δικέ μα πληροφορίε. Εκεί πρέπει να κεντρωθούμε. Ο κ. Μπουσίνη ανέφερε επίση την εμβληματική μα πολιτική, ε, δηλαδή κατά δίκη τη θανατική ποινή. Εμεί ε, καλούμε την ε, Σαουδική Αραβία, αν όχι να καταργήσει την θανατική αρχή, που είναι και η βασική μα προτεραιότητα, τουλάχιστον να υπάρξει ένα μορατόριο στι εκτελέσει, στι θανατικέ ποινέ και να προσπαθήσει να σεβαστεί τουλάχιστον προς εκτελέσει τα κατώτατα πρότυπα που θεσπίζουμε στις κατευθυντήριες γραμμές μας, ε, στις κατευθυντήριες γραμμές ECOSOFT. Ευχαριστώ. Thank you and... Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που με ενημερώσατε και για την ε, κατάσταση ό,τι αφορά την κατάσταση του κύριου Κασκάρη. Μιχάλης πληροφορίε ε, από που μου είχε γράψει ο κύριος Σούλτσε, τώρα είναι θετικά αυτά που λέτε. Ποιοι θέλουν το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριο Πρέσβή. Ακούστε κύριε Πρέσβη, πριν σα δώσω το λόγο, θα ήθελα πρώτα να ακούσουμε τα μέλη τη Επιτροπή μα. Μπορεί να θέλουν ερωτήσεις, να κάνουν ή να σχολιάσουν κάτι. Επειδή θεωρώ ότι είμαι και εγώ μέλος τη επιτροπή, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μπουσί. Πολύ καλό είναι αυτό που λέτε ότι έχετε διάλογο κτλ. Ε, υπάρχει μια σιωπηρή διπλωματία σε εξέλιξη. Είπατε ότι έχετε πετύχει κάποια θετικά αποτελέσματα σε ατομικές ε, υποθέσεις, όταν έχουμε δηλαδή καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, μην μας δώσετε ονόματα, απλά έχετε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό ήθελα να ξέρω. Well, I'm almost obliged to say yes. Ε, σχεδόν υποχρεωμένος να πω ναι. Και απαντάω ναι, γιατί πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ανοιχτός διάλογος, ακόμη και για ατομικές υποθέσεις, μπορεί να οδηγήσει αυτό σε θετικά αποτελέσματα. Και έχουμε κάποιες υποθέσεις, κάποιες περιπτώσεις. Εσείς μιλήσετε για σιωπηρή διπλωματία. Όχι ανοιχτή, δημοσιοποιημένη θα την χαρακτηρίζω Εδώ μπορούμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Είμαι αισιόδοξο ε, για τα αποτελέσματα που μπορεί να εγγυθεί αυτό ο συνεχής διάλογο που έχουμε με τι αρχέ τη Σαουδική Αραβίας, ακόμη και για μεμονωμένες ε, υποθέσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον πρέσβη κ. Φαϊσάλ. Αν δεν με πατά μου, είναι η πρώτη φορά που παρακολουθείτε τι συζητήσεις μας στην Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το ενδιαφέρον σας. Πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας πω ότι στην Επιτροπή μας έχουμε τον κανόνα ο πρέσβης όποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο να μπορεί να το κάνει, αλλά η παρέμβασή του περιορίζεται σε τρία λεπτά. Αν θέλετε να μας κάνετε μια περαιτέρω ανάλυση από τη δική σας πλευρά, να σας ακούσουμε ευχαρίστως, αλλά μπορείτε να μας στείλετε πιο αναλυτικά τις παρεμβάσεις εγγράφως. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε δεν είναι αρκετά τα τρία λεπτά, αλλά όπως είπατε έχουμε και την άλλη δυνατότητα Εγγράφω να σας παρουσιάσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο πιο αναλυτικά τις θέσεις μας. Καταρχάς ήθελα να πω ότι το βασίλειο της Σαουδική Αραβία είναι ένα κυρίαρχο ασλαμικό ε, κράτος. Το σύνταγμα του βασίζεται στην Ισλαμική πίστη και τη Σαρία, το Κοράνι και τις διδαχές του προφήτη Μωάμεθ. Βέβαια, ε, είμαστε υπέρ της ανοχής, ε, της δικαιοσύνης και η πίστη μας ζητεί ε, το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το άρθρο 26 του βασικού μας νόμου λέει ότι το κράτος προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με την Ισλαμική Σαρία. Για αυτό το σκοπό, κυρία Πρόεδρε, η χώρα μας, η Αραβία, προσχώρησε σε ορισμένες περιφερειακές και διεθνεί συνθήκες και συμβάσεις, την Διεθνή Σύμβαση για την εξάλληψη κάθε μορφή φιλετικής διάκριση, Σύμβαση για την εξάλληψη κάθε μορφής διάκριση κατά των γυναικών, τη Σύμβαση κατά των βασανισμών, βασανιστήριων και άλλη απάνθρωπης ή ε, ταπεινωτικής μεταχείρισης, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών, Ραβικό Χάρτη των Δικαιωμάτων, Διακήρυξη του Καΐρου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το χάρτο του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες συνθήκες. Εσωτερικά τώρα, το 2005, θεσπίσαμε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται για ένα κυβερνητικό φορέα που υπάγεται άμεσα στον Πρωθυπουργό, που είναι ο Βασιλέας φυσικά, και εξασφαλίζει την υλοποίηση ε, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους κρατικούς φορείς και έχει ε, την απόλυτη εξουσία για την επιθεώρηση και την παρακολούθηση των επιπέδων ε, των εργασιών όλων των κρατικών και μη κρατικών οργανισμών στη Σαουδική Αραβία. Το 2004 επίσης δημιουργήθηκε η Εθνική Εταιρεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από, μια ε, από ορισμένους ακτιβιστές, μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εργάζεται για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης και την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία φόντος συστάθηκε, εργάζεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με βάση, όπως είπα, την Ισλαμική Σαρία. Πρόσφατα μας κατηγόρησαν ως φονταμεταλιστές και τρομοκράτες. Those uh, uh, acts and especially the ideologies and the mindset behind. Υπάρχουν ε, δράσεις τέτοιες τις οποίες καταδικάζουμε και θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε. και έχουμε και δεχθεί και εμείς τέτοιες επιθέσεις. Ε, η Ισλαμική πίστη, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι τα περισσότερα δικαιώματα από οποιαδήποτε ε, αναφέρεται ήδη σε άλλες διακηρύξεις ή συνθήκες. Σήμερα οι γυναίκες στη χώρα μας είναι ισότιμοι εταίροι προς τους άνδρες, ε, ιδίως ό,τι αφορά την εργασία, την εκπαίδευση και τα βασικά δικαιώματα. Ε, στο Συμβούλιο Σώρα ο Βασιλέας ε, Αμπτούλαχ ε, έχει συμπεριλάβει γυναίκες που είναι μια διεθνής κοινοβουλευτική ένωση. Οι γυναίκες επίσης έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιες και να ψηφίζουν και να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Ολοκληρώνοντας, σε αναγνώριση από την κοινότητα του έργου και των προσπαθειών της Σαουδικής Αραβίας ε, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Σαουδική Αραβία είναι μέλος ε, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ από το 2005 και επανεκλεγήκαμε για τρίτη φορά. Σας ευχαριστώ. Thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Εάν το επιθυμείτε, και εμένα θα με ενδιαφέρει να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή τις αλλαγές που, στις οποίες έχετε προβεί την υπογραφή συνθήκων και τις επιφυλάξεις που έχει κάνει η κυβέρνησή σας για ορισμένες συνθήκες όσον αφορά το περιεχόμενό τους, όσον αφορά επίσης τη συνθήκη για το καθεστώς των γυναικών. Θα μπορούσατε να μας στείλετε εγγράφος ή κάποια έκθεση ε, και για την ιστοσελίδα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την οποία έχετε προβλήματα. Θα ζητήσω τώρα από τον κύριο και να συνοψίσει τη συζήτηση και μόλις ε, έλεγξα στο κοινοβούλιο μας ε, ψηφίσαμε ένα ψήφισμα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Δικαιραβία το Δεκέμβριο του 2007 επίγον ψήφισμα εστιαζόμενο στα δικαιώματα των γυναικών. Πιστεύω ότι θα πρέπει Επίσης, ε, να δούμε τα όσα μας παρουσίασε ο κύριος Βουίλκε και τις πολύπλευρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, αλλά τονίσαμε επίσης ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια προσέγγιση εστιασμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τις συζητήσεις μας με τη Σαουδική Αραβία. Θα ήθελα λοιπόν οι πολιτικές ομάδες να εξετάσουν μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να ε, συνταχθούν και να συντάξουν ένα νέο ψήφισμα προς υποστήριξη των εξελίξεων στη Σαουδική Αραβία αλλά και προς υποστήριξη του έργου της αντιπροσωπείας ε, των Ηνωμένων Εθνών επιτόπου. Κύριε Βίλκε, παρακαλώ, έχετε τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπασίνη, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Και ευχαριστώ κύριε Αλεξανδρίδη ε, για τα σχόλιά σας. Μερικές φορές νιώθω περίεργα όταν προσπαθώ να περιγράψω διεθνείς ε, ε, κατηγορίες εναντίον κυβερνήσεων και της Σαουδικής Αραβίας και τις συγκρίνω με τις συχνές κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Υπουργείων Εξωτερικών διαφόρων χωρών προς άλλες χώρες. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε έναν ιδιωτικό διάλογο, αλλά όπως ε, ε, τονίσαμε θα πρέπει να δείξετε και αποτελέσματα. Όταν μιλάτε με φίλους, τότε αναμένετε οι φίλοι σας να σας παίρνουν στο σοβαρά και νομίζω ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα με, τις, με τη Σαουδική Αραβία. Το Κοινοβούλιο πιστεύω έχει κάνει μια δήλωση όσον αφορά τη σύλληψη ορισμένων χριστιανών ε, κατοίκων Αιθιοπίας, ε, υπηκών της Αιθιοπίας που έχουν το δικαίωμα να συγκεντρωθούν για θρησκευτικούς σκοπούς σε έναν ιδιωτικό οίκο και αυτοί συλλήφθηκαν και από ό,τι ενημερώθηκα παραμένουν σε κράτηση παρά τις διαφορές διαμαρτυρίες όσον αφορά το ζήτημα του Χαμσακασκάρη έχω διαφορετικές πληροφορίες από εσάς εσείς ίσως να έχετε πιο νέες, εγώ έχω πριν από μια εβδομάδα, βρίσκεται σε απομόνωση, κρατείται σε απομόνωση, δεν έχει πρόσβαση σε νομική υποστήριξη, δεν έχει παραπεμφθεί η υπόθεση του στην εισαγγελία, συνεπώς ε, βάσει του νόμου της Σαουδικής Αραβίας δεν υπάρχει νομική βάση για την κράτησή του. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει μια λύση για αυτή την περίπτωση, ίσως αυτό να συμβαίνει. και ίσως να προσπαθεί να βρει μια λύση σιωπώντας τον για να μην διαταράσει ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας όσον αφορά τη θανατική ποινή αποτελεί ζήτημα που μας ανησυχεί η Σαουδική Αραβία καταψηφίζει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για τα η θανατική ποινή λέγοντας ότι αντιδεχτεί στην Σαρία υπάρχει αυτή η θανατική ποινή για την κατανάλωση και διακίνηση ναρκωτικών. Είναι από του ελάχιστου κωδικοποιημένου νόμου τη Σαουδική Αραβία. Θα πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση τη Σαουδική Αραβία μήπω μπορεί να ρίξει μια δεύτερη ματιά για τη θανατική ποινή για τη διακίνηση ναρκωτικών. Κατά πόσο υπάρχει κάποια ένδειξη ότι έχει αποτρεπτικά αποτελέσματα. Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Έχω μιλήσει με κρατουμένου που έχουν κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών. Ορισμένοι ε, θανατοπινίτες οι οποίοι βασανίστηκαν για να υπέστησαν βασανιστήρια για να ομολογήσουν. Μια τρομακτική ιδέα να βασανίζεις κάποιον ε, για να ομολογήσει πριν ε, υποστεί την θανατική ποινή. Τώρα οι εκτελέσεις δεν γίνονται σε δημόσιες πλατείες όπως γινόταν παλιά, αλλά εντός των φυλακών και αυτό μας ανησυχεί, διότι ελάχιστες εκτελέσεις δημοσιοποιούνται. Η Σαουδική Αραβία δεν κοινοποιεί σε θανατοπινίτες το γεγονός ότι θα πρέπει να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους. Ο νόμος, ε, ο αντιτρομοκρατικός νόμος, όπως υποτίθεται ότι αναθεωρεί, αναθεωρήθηκε, εισήγαγε πάνω από 30 νέα εγκλήματα, μη βία τα οποία εφίστανται τη θανατική ποινή. Θα πρέπει να καταργηθούν αυτές ε, οι περιπτώσεις θανατικής για μη βία εγκλήματα. Αυτά είχα να πω για τα διάφορα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν. Ε, επίσης προσδοκώ την αξιολόγηση των τεσσάρων ετών μετά από την ε, παγκόσμια περιοδική αναθεώρηση και την υλοποίηση των συστάσεων. Η Human Rights Watch έχει απαγορευτεί να επισκεφθεί τη χώρα. Έχουμε γράψει την Επιτροπή που αναφέρατε ζητώντας πρόσβαση στη χώρα χωρίς να λάβουμε ποτέ καμία απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πιστεύω ότι τώρα όλοι γνωρίζουμε κάπως περισσότερα για την κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Έχω λάβει μια επιπλέον πληροφορία ότι στο δεύτερο γύρο της παγκόσμιας περιοδικής αναθεώρησης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να υποβάλει μια έκθεση τον Οκτώβριο του 2013. Ως ε, πρόεδρος εδώ της Επιτροπής, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε από τώρα μέχρι εκείνη τη στιγμή το 2013 για το τι είδο υποστήριξη θα μπορέσουμε να παρέχουμε ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Ευχαριστώ κύριε Βουλκέ. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Έχουμε την πρώτη εξέταση για, για την, το σχέδιο σύστασης σε ό,τι αφορά τον ειδικό αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο εισηγητής του Κοινοβουλίου, η εισηγητρία είναι η κυρία Αντρικίνα. Στις 26 Απριλίου έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή μας, επειδή το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχουν δώσει ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Σα υπενθυμίσω ότι και εμείς ε, θα ακολουθήσουμε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά τον διορισμό του ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον Ιούνιο στα πλαίσια του πακέτου αναθεώρησης. Να πω και το εξής, η κυρία Αντρικίνα ζήτησε από όλες τις πολιτικές ομάδες και από τους κοιόδης να προβούν σε συστάσεις ως προς το σχέδιο αυτό. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τυρκουάς εβδομάδα. Θα θέλετε λοιπόν να μας ενημερώσετε για το πώς έχει η κατάσταση και πώς ε, έχουν εξελιχθεί οι συζητήσεις και μετά θα πω δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Αντρικένε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έγινε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων στις 26 Απριλίου. Και το πρώτο σχέδιο διανεμήθη στους συντονιστές από όλες τις πολιτικές ομάδες. Προθεσμία για τις προτάσεις ήταν η προηγούμενη Παρασκευή και ευχαριστώ την κυρία Μπάρμπαρα Λοχμπίλτερ για την, ε, Λοχμπίλερ για τη συμμετοχή της. Έχουμε ήδη εντάξει κάποιες από τις προτάσεις σας ε, στο σχέδιο το οποίο ε, διανεμείται στους, διανεμείται στους Στο μέλλον ενδεχομένως να δεχτούμε προφορικές τροπολογίες σύμφωνα με τον κανονισμό 22 Μαΐου είναι η προθεσμία για την κατάθεση προφορικών τροπολογιών, γιατί 24 Μαΐου θα το κοιτάξουμε το θέμα στην εβδομάδα του Στρασβούργου. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μας πει το Συμβούλιο και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, γιατί αν δεν υπάρχει καταπήγον χαρακτήρας για το πακέτο ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αν υπάρξει σχετική αναβολή στο Συμβούλιο, αυτό θα σημαίνει ότι έχουμε πιο πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πρωτού ε, ψηφίσουμε το σχέδιο αυτό. Τα βασικά ζητήματα έχουν ήδη παρουσιαστεί στις 26 Απριλίου. Οι βασικές ιδέες λοιπόν είναι οι εξής ενώ ο διορισμός του ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί επισήμως απόφαση του Συμβουλίου και χρειάζεται ειδική πλειοψηφία για το διορισμό του ειδικού αυτού αντιπροσώπου και η απόφαση αυτή βασίζεται σε πρόταση της ύπατης ε, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ο ειδικό ε, αντιπρόσωπος θα πρέπει να μιλάει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο εξ ονόματος του Συμβουλίου ή της Επιτροπής ή του ειδικού αντιπροσώπου. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η διαφάνεια της θέσης αυτής, προτείνουμε μία ανταλλαγή απόψεων σε συναντήσεις κυκλισμένων των θηρεών της Επιτροπής ε, Κοινής, συνεδριάσεις κοινές της Επιτροπής ε, ε, εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Προτού γίνει η ψηφοφορία στο Συμβούλιο και όχι όπως προτείνεται στο σχέδιο να λάβουμε από την Υπηρεσία εξωτερική Δράσης πληροφορίες μετά το διορισμό και πριν την ανάληψη των καθηκόντων από τον ειδικό αντιπρόσωπο. στο σχέδιο σύστασης μιλάμε για τους πολιτικούς στόχους. Τι θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε. Να βελτιωθεί η συνοχή και η προβολή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε ο ειδικό αντιπρόσωπος να είναι ε, υψηλού επίπεδου ομόλογος των ε, αντίστοιχων αξιωματούχων σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμών σε οργανισμούς και να μπορεί να συμμετέχει και στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, αλλά και σε περιφερειακές σχετικές οργανώσεις. Επίσης, προτείνουμε ο ειδικό αντιπρόσωπος να ηγείται συζητήσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να είναι υπεύθυνο για τι διαπραγματεύσει με τρίτε χώρε. Σε ό,τι αφορά την εντολή τώρα του ειδικού αντιπροσώπου, λαμβάνοντα υπόψη ότι πρόκειται να ενεργεί υπό την αιγίδα της ύπατης αντιπροσώπου, προτείνουμε να έχει ισχυρή ανεξάρτητη εντολή χωρίς ειδικές, ειδικούς θεματικούς περιορισμούς να μπορεί να δρά γρήγορα και αποτελεσματικά. Επίσης, στο σχέδιο σύστασης αναφέρουμε ότι η εντολή θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές που διέπουν ε, τις πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρουμε ότι ο δικός αντιπρόσωπος θα πρέπει να έχει ασφαλώς τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες, εμπειρία, ε, πείρα στον τομέα των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διάρκεια της θητείας, προτείνουμε να διορίζεται για δύο έως δυόμιση έτη για να υπάρχει συνέχεια και να είναι ανανεώσιμη άπαξ η θητεία του. Επίσης αναφέρουμε ότι ο ειδικό αντιπρόσωπος θα πρέπει να εργάζεται, να συνεργάζεται στενά με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, με τους εμπειρογνώμονες αλλά και με διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν αποτελεί το περιεχόμενο του σχεδίου μας. Να κλείσω λέγοντας ότι προτείνουμε μάλλον ότι ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τον διορισμό του δικού αντιπροσωπού για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2009. Και το 2010 ξαναφέρθηκε η πρόταση αυτή, η οποία επιπλέον, επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά. Και περιμένω την, προσπα... την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων. Αν θέλουμε να είναι αποτελεσματικός ο τρόπος δράσης και να δρά με συνοχή, προκειμένου να είναι σωστή η πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι πολύ απαραίτητο το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Ντόνσκινς. Ευχαριστώ πολύ. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή μου προς την συνάδελφο Αντρική και αυτά που είπε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πρωτοβουλία της ALDE. Αφορά μια επιστολή που στείλαμε στην Βαρόνη Κάθριν Άστον. Την υπογράφει ο Γκί Φερχόφστατ, ο κύριος Μακμίλαν Σκότ και εγώ, ο υποφαινόμενος. Εκεί υπογραμμίζουμε τη σημασία τις θέσει του ειδικού αντιπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στηρίζουμε την ιδέα αυτή. Δεν θέλω να σα ε, διαβάσω ή να επαναλάβω λέξη προ λέξη την επιστολή, αλλά να σα ενημερώσω για δύο-τρία πράγματα. Να τονίσω ότι λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερο σε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διατρέχουν όλη την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να οριστεί ο ειδικό αντιπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο να τονιστεί η προβολή, ο αντίκτυπος της πολιτικής ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεκτικότητα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εφαρμοστεί το πακέτο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ΕΦΕΣΥ πριν από το καλοκαίρι και επίσης να, υπάρχει, να εφαρμοστεί και η δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σχέδιο δράσης. Τέλος, ο ειδικός αντιπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να έχει ένα διεθνές προφίλ, να διαθέτει εμπειρία, αποδεδειγμένη αφοσίωση στην υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια επιτυχημένη τέτοια θέση θα πρέπει να ανατεθεί ε, σε μια γνωστή προσωπικότητα, ε, σε έναν που θα γνωρίζει το διεθνές δίκαιο, θα έχει αρκετές επιστημονικές γνώσεις ώστε να μπορεί και να συνεργαστεί με διεθνείς ομολόγους. Επίσης, ε, ζητούμε τη συλλογικότητα, να εγκριθεί δηλαδή από όλες τις πολιτικές ομάδες, γιατί όλοι προς την ίδια κατεύθυνση εργαζόμαστε. Την υπογράφει, παραλαμβάνω, την επιστολή, ο Φερχόφστατ, ο Άντρου Μακμίλαν Σκότ, εγώ και μετά λέμε με εκτίμηση στο τέλος. Δεν νομίζω ότι στον επιστολή σας υπάρχει κάτι αντίθετο με τις προτάσεις μας, έτσι σας το λέω ενημερωτικά. Ναι, πράγματι. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη. Υπάρχουν κάποιες άλλες δραστηριότητες, κάποιες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε ε, επιπροσθέτως, αλλά την ίδια φωνή, ε, την ίδια γλώσσα μιλάμε όλοι. Κύριο Σταβάρης, ευχαριστώ πολύ. Αν δεν σας πειράζει θα μιλήσω πορτογαλικά. Σας δίνω λίγα δευτερόλεπτα. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγητριά μας, την κυρία Αντρικίνε. Και εμείς πιστεύουμε ότι μεγάλο μέρος των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί ε, στην Υποεπιτροπή των Δικαιωμάτων ή σε διμερές επαφές και συνομιλίες έχουν ληφθεί υπόψη σε μεγάλο βαθμό. Είναι λοιπόν σε αυτό το στάδιο σημαντικό να ενισχύσουμε ακριβώ τι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάπου να αναφέρουμε κάποιους προβληματισμούς και σε κάποια άλλα σημεία να διευκρινίσουμε κάπως περισσότερο τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία. Συμφωνώ με όλα όσα είπε ο προλαλής σας κύριος Ντόνσκης. Όλοι είμαστε ενθουσιώδεις απέναντι στην δημιουργία της νέας θέσης αυτής, ενός ειδικού αντιπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι έχει σταθμίσει το Κοινοβούλιο τα υπέρ και τα κατά της δημιουργίας της θέσης αυτής. Είπαμε ήδη ότι δεν θα θέλαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να γκαιτοποιηθούν, να περιοριστούν δηλαδή σε ένα κομμάτι μόνο τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτω, θέλουμε να είναι στο επίκεντρο τη Ευρωπαϊκή Εξωτερική πολιτική. για να εγγυηθούμε την διασύνδεση μεταξύ τη εξωτερική πολιτική και τη εσωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δοθεί έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα και στα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν ή όλα θα εξαρτηθούν από το προφίλ του ανθρώπου που θα αναλάβει τη θέση αυτή πρέπει να φροντίσουμε να είναι κάποιος ή κάποια με έντονα την προσωπικότητα που θα είναι ειλικρινής, τίμιος στον τρόπο τον οποίο θα απευθύνεται και στην ε, κοινότητα των πολιτών και στους διάφορους θεσμούς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο αφού εμείς είμαστε ε, το Δημοκρατικό Όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό στηρίζω την πρόταση της έκθεσης της κυρίας Αντρική, δηλαδή ο αντιπρόσωπος πριν το διορισμό του να παραστεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής μας γιατί είναι σημαντικό να ακούσουμε τι θα έχει να μας πει το εν λόγω άτομο για το έργο το οποίο θα επιτελεί. Να δούμε ποιο είναι το ιστορικό του, ποιε είναι οι επιδόσεις του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμφωνώ με τις γενικές συστάσεις για το προφίλ του ατόμου αυτού. Κάτι άλλο σημαντικό θα πρέπει το άτομο αυτό να έχει στη διάθεσή του δυνατότητες μέσα για να φέρει σε πέρα στο έργο του. Πρέπει να πάμε πιο μακριά από όσα περιλαμβάνονται στην αναφορά της κυρίας, στην έκθεση της κυρίας Θα πρέπει ο δικός αντιπρόσωπος να έχει στη θέση του να πάρει τεχνική εμπειρία, να συνεπικουρείται από άτομα που θα είναι σύνδεσμοι με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, που θα συλλέγουν πληροφορίες, γιατί πολύ συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνουμε ότι είναι δύσκολο να συλλεγούν αξιόπιστες πληροφορίες. Πολλές φορές ε, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας δίνουν αντιφατικές πληροφορίες. Το γραφείο του δικού αντιπροσώπου, αν και δεν θέλουμε να τα κάνει όλα, βέβαια, γιατί δεν μπορεί κανείς να τα κάνει όλα, Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να, ε, παρόλα αυτά να ενισχύσει την ε, προβολή και την αποτελεσματικότητα της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα. Να μην λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα, να λέμε ότι πρέπει να αγγιηθούμε τη συνεκτικότητα. Και μόνο έτσι θα ενισχύσουμε την ορατότητα, την προβολή. Συνεκτικότητα λοιπόν, συνέπεια εσωτερικής εξωτερικής πολιτικής. εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας ε, και του πολίτη. Στην παράγραφο 1, στο ε, υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αποστολές. Ο ειδικός αντιπρόσωπος δεν θα πρέπει μόνο να, να πραγματεύεται αυτά τα οριζόντια θέματα, αλλά θα διατυπώνει και συστάσεις. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, ε, διατύπωση συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλες προσθήκες. Είναι ήδη μακρύς ο κατάλογος, αλλά όλα όσα περιλαμβάνει είναι σημαντικά. Υπάρχει μια σειρά αποστολών που θα αναλάβει ο ειδικός αντιπρόσωπος. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε λοιπόν το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση των βασανιστήριων, βασανισμών, καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Ελευθερία έκφρασης ε, και θρησκευτική ελευθερία, προστασία παιδιού κτλ. Νομίζω ότι λείπει η καταπολέμηση των διακρίσεων, που είναι και το ουσιώδες. Είτε σε συνάρτηση με το φύλλο, είτε για θρησκευτικού λόγους, διάκριση ανδρών γενικών και ούτω καθεξής. Στο λατινικό «αι» εδάφιο της παραγράφου αυτής, θέλω να διευκρινιστεί το εξής. Όταν λέμε ότι θα πρέπει να συνεισφέρει στην ενσωμάτωση διάσταση του φύλου, σε, του μάλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όλες τις πολιτικές και σε όλα τα θεσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, με συμφωνώ με τη γενική αυτή ε, διατύπωση. Αλλά όταν λέμε σε όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, σε αυτά τα θεσμικά όργανα περιλαμβάνεται και το Ευρωκοινοβούλιο. Μήπω θα έπρεπε να διευκρινίσουμε για ποια θεσμικά όργανα γίνεται λόγο. Μιλάμε μόνο για συμβούλια και Κομισιόν ή συμπεριλαμβάνεται και το Ευρωκοινοβούλιο. Και θα πρέπει να πείτε τι συστάσει πρέπει να διατυπωθούν για το Κοινοβούλιο. Γιατί το λέω αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνο σύγχυση. και γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια. Στο εδάφιο J, λατινικό, όπως είπα και πριν, λέμε ότι ο εκπρόσωπος, ο ειδικός αντιπρόσωπος θα πρέπει να αναφέρεται τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Πέραν αυτή τη έκθεση και αναφορά προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώ εξελίσσεται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, ειδικό αντιπρόσωπο θα πρέπει επίση τακτικά να μα λέει τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει. Δηλαδή, δεν έχει μόνο υποχρέωση ενημέρωση, θα πρέπει να έχει και υποχρέωση υλοποίηση. δηλαδή να μα υποβάλει μέτρα. Αυτά έχω να πω. Να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς την εισηγήτρια που εργάστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Σας στηρίζουμε και η ομάδα μου και εγώ προσωπικά, ώστε οι στάσεις σας να έρθουν σε αίσιο πέρας και να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βέβαια να εισακουστούν και από τους άλλους, τα άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. Μετά τον κύριο Υπάρχει κάποιος άλλος? Όχι, μετά από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λειτουργούμε με την ταχύτητα του φωτός εδώ, συνεπώς πρέπει να έχουμε ταχύτητα της αντιδράσεις. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ τον κύριο Σαντροκιανέ για το σχέδιο εγγράφου για το σχέδιο συστάσεων που μας παρουσιάσατε. Πιστεύω ότι είναι ένα εξαιρετικό έγγραφο ύψης της ποιότητας. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να συμπληρωθεί με μερικά στοιχεία, διότι είμαι βέβαιος ότι όλοι θεωρούμε ε, τον ειδικό αντιπρόσωπο ως κάτι διαφορετικό. Έχουμε την τάση να φορτώνουμε αυτό το συγκεκριμένο άτομο με υπερβολικά πολλές ευθύνες πριν το πράξουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό το άτομο θα μπορέσει να φέρει εις πέρας όλα αυτά τα καθήκοντα. Δεν πρέπει λοιπόν να υπερφορτώνουμε ε, τον ειδικό εκπρόσωπο με το πώς φανταζόμαστε εμείς ότι ε, θα έπρεπε να είναι τα καθήκοντά του. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι το λόγο άτομο θα δρά με, σε κάποια επίπεδα δομής ε, της συνθήκης, ε, των συνθήκων γενικότερα και το καθεξής. Αυτό που λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε πρώτα. Επικροτώ το σχέδιο εγγράφου της κυρίας Αντρικένε. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά φιλόδοξο. Είμαστε εμεί φιλόδοξοι και αναμένουμε πολλά από τον ή την υποψήφιο που θα επιτελέσει αυτές τις λειτουργίες. Θα θέλαμε το εν λόγω άτομο να έχει κάποιο πρεστής, Χαρί στη δική του ή της εμπειρία, το παρελθόν, την εκπαίδευση. Έχουμε πολλά παραδείγματα θεσμών που δημιουργούμε από τους οποίους έχουμε τεράστιες προσδοκίες. Ενώ το άτομο που καμιά φορά καλύπτει ένα συγκεκριμένο πόστο είναι πολύ δεν είναι επαρκές για να καλύψει το συγκεκριμένα καθήκοντα. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε το σωστό άτομο για τα συγκεκριμένη θέση και πιστεύω ότι επίση είναι εξαιρετικά σημαντικό εδώ να εγκαθιδρύσουμε μια σωστή σχέση μεταξύ αυτής της νέας θέσης και αυτού του νέου ατόμου που θα την καλύψει τη σχέση μεταξύ αυτού του ατόμου και της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Φυσικά θέλουμε να έχουμε σωστές αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες γωνιές της γης. Ορισμένες φορές υπάρχουν αμφιβολίες. Έχουμε αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. Μπορούμε λοιπόν ορισμένες φορές να επαληθεύσουμε μέσω της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ή μέσω των αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πόσο οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι σωστές ή όχι. Επίσης Έχουμε μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, που επίση μπορούν να αποτελέσουν την πηγή σχετικών ε, αξιόπιστων δεδομένων σε σχέση με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω όσον αφορά το ζήτημα και τη σπουδαιότητα του δημοσιολαβητή. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ρόλος. Έχουμε δημοσιολαβητή για τα κράτη-μέλη ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε τρίτα κράτη ε, μερικές φορές φυσικά δεν είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι από τη δομή αυτή ε, της, θέση αυτής της θέσης του δημοσιολαβητή της απόσπασης δημοσιολαβητών σε άλλες χώρες αλλά σε, στις χώρες όπου υπάρχει δημοσιολαβητής πιστεύω θα πρέπει να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το δίκτυο. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Πολλές φορές ακούγεται στις συζητήσεις μας ότι έχουμε παρατηρήσει πως ορισμένες οδηγίες, ορισμένοι κανόνες που προσπαθούμε να επιβάλλουμε από ψηλά απλά δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Δεν τις ακούει κανένας. Αν όμως χώρες έχουν καλές πρακτικές και τις ανταλλάσσουν, αυτό αποτελεί μια εξαιρετική σύσταση, εξαιρετική ενθάρρυνση για τις χώρες που ξεκινούν τη διαδρομή της προς τη δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε περάσει ήδη στο τέλος